για να έχουμε ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Ντάνσερ, ε, ο οποίος θα μας παρουσιάσει το πρόγραμμα του οργανισμού το πρόγραμμα εργασίας του ΕΚΑ, το θέμα των φόρων των που επιβάλλονται, πώς έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα, γιατί πρόσφατα μια αντιπροσωπεία από το Κοινοβούλιο επισκέφθηκε τον ΕΚΑ. Μπορέσαμε να συζητήσουμε μαζί τους. Ήταν πολύ ενδιαφέρον το πρόγραμμα της επίσκεψης και ο κύριος Ντάνσετ μαζί με τους συναδέλφους του μας ε, παρουσίασε μια επισκόπηση του τι κάνουν. Θα έλεγα λοιπόν να ξεκινήσουμε το σημείο αυτό, να δώσουμε το λόγο στον κύριο Ντάνσετ και μετά η κυρία Χάση που είναι υπεύθυνη για τις επικοινωνίες μας με τον ΕΚΑ και φροντίζει να παραμένει στενή η σχέση μας με αυτόν τον οργανισμό. Θα κάνει τα δικά της σχόλια και θα ακούσουμε και τους υπόλοιπους συναδέλφους. Κύριε Ντάνσετ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, Αντιπρόεδρε, μέλη της Επιτροπής, είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι μαζί σας σήμερα και πάλι για να σας φέρω νέα από τον Οργανισμό για τις Χημικές Ουσίες, το χιονισμένο Ελσίνκι. Θα σταθώ σε κάποια από τα επιτεύγματα που πετύχαμε από την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε, αλλά περισσότερο θα μιλήσω για τις φιλοδοξίες μας για την προσεχή έτη. Έπειτα θα έχουμε και πολύ χρόνο για να ακούσω τις δικές σας ερωτήσεις και να τις απαντήσω. Δεν σας φαίνεται ότι ο χρόνος τρέχει Πραγματικά δεν φαίνεται να έχει περάσει πολύ καιρό από τότε που σα μιλούσα για τα μεγάλα επιτεύγματα τη πρώτη προθεσμία που είχαμε για την πρώτη φάση του ΡΙΤΣ. Φέτο βεβαίω αναμένουμε τη δεύτερη προθεσμία για τον Μάιο, να λήξει για τον Μάιο του 2013. Όλε μα οι προετοιμασίε αφορούν την καθοδήγηση και τα εργαλεία πληροφορική και έχουν περατωθεί, καθώ ε, ξεκινάει από αύριο ένα εξάμεινο μορατόριο. Η καταγραφή θα είναι κάτι που θα το δει η ομάδα των ε, υπευθύνων επαφών και των ενδιαφερομένων του μηχανικού κλάδου. Ω προ την ε, αποτίμηση, νομίζω ότι πετύχαμε την καταλεκτική ημερομηνία του Νοεμβρίου για την ε, αξιολόγηση των προτάσεων δοκιμών, όπως πρέβλεπε η πρώτη προθεσμία. Έχουμε ήδη μια νέα στοχευμένη στρατηγική για να έχουν μεγαλύτερο επίπεδο φακέλων καταγραφή συμμόρφωσης και για να δούμε κατά πόσον θα έχουμε και τις, ανάλογε τις ανάλογες αποφάσεις ελέγχου. Επίσης θα πρέπει να επιτελεστεί πρόοδος ε, στις ουσίες ε, σε νάνομορφές και να ληφθούν οι πρώτες σχετικές αποφάσεις. Επίσης υπάρχουν ακόμη πολλές ουσίες που μας ενδιαφέρουν στον κατάλογο με τις υποψήφιες ουσίες. Ελπίζω θα πετύχουμε το φιλόδοξο στόχο που έχει θέσει ο Αντιπρόεδρος Ταγιάννη και ο Επίτροπος Ποτότσνικ από το 2010, ώστε να φτάσουμε τις 136 ουσίες στον κατάλογο μέχρι το τέλος της χρονιάς. Ω προ την ε, διάδοση και την προβολή, έχουμε επίση επιτελέσει σοβαρή πρόοδο και αυτή την εβδομάδα δημοσιεύουμε τα ονόματα των εταιριών που έχουν ε, καταγεγραμμένε ε, ουσίε στον ιστότοπό μα. Επίση, ολοκληρώνουμε την αποτίμηση των αιτήσεων απορρίτου που έχουν υποβληθεί βάσει τη πρώτη προθεσμία για την πρώτη καταγραφή. Θα μιλήσω αργότερα για τα διοκτώνα και τι σχετικέ προετοιμασίε. Τώρα θα ήθελα να σα μιλήσω για τι φιλοδοξίε μα για το μέλλον. Τι εννοώ λέγοντας φιλοδοξία. Το λεξικό ορίζει τη φιλοδοξία ως μια ισχυρή επιθυμία και από αποφασιστικότητα για επιτυχία. Επίσης, ένα φιλόδοξο εγχείρημα ορίζεται ως ένα εγχείρημα με υψηλές προσδοκίες, δύσκολο όμως να πετύχει κανείς. Στην ΕΚΑ εμείς ε, νομίζω ότι αποδεικνύουμε το διτό νόημα της λέξης φιλοδοξία και το επιδιώκουμε. Ε, έχουμε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα εργασίας με ανάλογους στόχους. το όραμά μας είναι να γίνουμε η πρώτη αρχή παγκοσμίως, ρυθμιστική αρχή για την ασφάλεια των χημικών ουσιών, με τους φιλόδοξους στόχους του κανονισμού REACH και όπως μας ανέθεσαν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, όντως καλό είναι να έχουμε τέτοιους φιλόδοξους στόχους. Θα ήθελα να επισημάνω τρεις από τις πιο συγκεκριμένε φιλοδοξίες μας. Να ε, είμαστε περισσότερο ανεξάρτητοι, να φτάσουμε το ευρύτερο κοινό και να μα ακούει το κοινό με ε, περισσότερο ε, εύληπτες πληροφορίες και να συνεργαστούμε ακόμη πιο στενά με τους ε, ενδιαφερομένους και εταίρους. Η πρώτη μας από, φιλοδοξία αφορά την ανεξαρτησία μας και την ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων. Από τη στιγμή της ίδρυσής μας αυτό υπήρξε ο θεμελιός λήθος των εργασιών μας. Κάθε απόφαση που λαμβάνουμε πρέπει να βασίζεται σε επιστημονικές γνώσεις προκειμένου να λάβουμε ρυθμιστικές αποφάσεις και να έχουμε και βεβαιότητα για τις γνώσεις αυτές. Δεν θα πρέπει όμως να είναι μόνο ανεξάρτητες αυτέ οι γνώσει, αλλά θα πρέπει ω τέτοιε και να αντιμετωπίζονται. Από πέρσι έχουμε ανανεώσει την στρατηγική μα και την πολιτική για την ανεξαρτησία και προκειμένου να αποφεύγουμε συγκρούσει συμφερόντων. Είδατε την έκθεση από το ελεγκτικό συνέδριο φέτο, όπου αναφέρει κάποιου τομεί όπου θα μπορούσε να επιτελεστεί βελτίωση για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενε συγκρούσεις συμφερόντων. Πράγματι, οι απόψει του συγκλίνουν με τις δικές μας και σε πολλέ περιπτώσει συμπίπτουν, διότι η δημοσίευση τη έκθεση. Καθυστέρησε μεν, αλλά οι περισσότερε από τι συστάσει του είχαν ήδη εφαρμοστεί προτού δημοσιευτεί η έκθεση. Έχουμε υπόψη ότι για του Ευρωπαίου πολίτε ένα θεσμικό όργανο τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ισότιμο με κάποιο άλλο. Οπότε αν ε, πλήττεται η φήμη του ενό, αυτό βλάπτει όλου μα. Κάνουμε λοιπόν ό,τι μπορούμε προκειμένου ο ΕΚΑ να μην απογοητεύσει την ευρωπαϊκή οικογένεια, ούτε και τον εαυτό του. Η δεύτερη φιλοδοξία μας είναι να, μας, να είμαστε πιο ορατοί στο ευρύτερο κοινό. Το, ο ισότοπος του ΕΚΑ ήδη περιέχει πολλές πληροφορίες για χημικές ουσίες περισσότερε από οποιονδήποτε στον κόσμο. Θέλουμε να υπάρχει εύκολη πρόσβαση και να είναι χρήσιμε για του ενδιαφερομένου οι πληροφορίε αυτέ. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε τεχνική φύση πληροφορίε και σκοπό είναι να βελτιωθεί και η διαπαφή όπω υπάρχει στο διαδίκτυο, οι πληροφορίε αυτές πραγματικά να μπορούν να αξιοποιηθούν από τον καθένα. Και οι ενδιαφερόμενοι θέλουμε να μπορούν να βρίσκουν αυτά που αναζητούν όταν απευθύνονται στον ιστοτοπό μας. Η απλούστευση επίσης είναι πολύ σημαντικά για τις επόμενες καταγραφές που θα γίνουν βάσει της ε, προθεσμίας που έχουμε για το χρόνο, ακόμα και για εταιρείες που είναι περισσότερο άπειρες, οι οποίες θα είναι πιο πολλές. Χρειαζόμαστε απλές, σαφείς και στοχευμένες πληροφορίες στον ιστότοπό μας και για τις ουσίες που αναφέρονται και παράγονται. Θα πρέπει λοιπόν να συνεργαζόμαστε με το δίκτυο ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και του πιστοποιημένου ενδιαφερομένους για να βοηθήσουμε αυτέ τι μικρότερε εταιρείε. Η τρίτη μα φιλοδοξία είναι να συνεργαζόμαστε όλο και στενότερα με του ενδιαφερομένου. Από την αρχή της λειτουργίας μας οι ενδιαφερόμενοι έχουν συμμετάσχει στις εργασίες μας και πιστεύουμε ότι έχουμε μια καλή φήμη για το ανοιχτό πνεύμα που δείχνουμε. Οι ενδιαφερόμενοι αυτοί ε, συμμετέχουν στην διαδικασία λήψης αποφάσεων και στους ε, σχετικούς φορείς, στις εκδηλώσεις των ομάδων εργασίας και σε πολλές από τις δράσεις μας. Στην ε, πρώτη φάση λειτουργίας του, του ΡΙΤΣ, ο ΕΚΑ συνεργάστηκε στενά με τους ε, ενδιαφερομένους από τη βιομηχανία, προκειμένου να έχουμε εργαλεία και πρακτικές και πληροφορικής, αλλά και χρήσιμες φιλικές προς το χρήστη, ώστε να μπορέσουν οι εταιρείε να συμμορφωθούν επιτυχημένα με τους ε, σχετικούς νόμους. Βέβαια κάποιοι είπαν ότι ο ΕΚΑ είναι προκατελημένο υπέρ το μηχανικό του κλάδου, αλλά αυτό δεν είναι καθόλου ε, πραγματικό. Διότι θα πρέπει να διορθώσουμε αυτή την προκατάληψη, δείχνοντας ότι οι αιτήσει συναντήσεις μας με τους ε, ενδιαφερομένους ε, των πιστοποιημένων, με τους πιστοποιημένους ενδιαφερομένους και τους ενώσεις τους επιτρέπουν να καταρτήσουμε κοινού στόχους, στρατηγικού στόχους με τις αρμόδιες επιστημονικές ε, επιτροπές. Επίσης ε, έχουμε και περιβαλλοντικές οργανώσεις επιστοποιημένων ε, ενδιαφερομένων και η ανάλυση τους κάποιες φορές είναι, βασίζεται σε παρανοήσεις. Γι' αυτό φροντίζουμε να έχουμε επικοδομητικές συστάσεις και αυτές να αποφούνται στις εκθέσεις τους. Εν τω μεταξύ ε, έχουμε άτυπο διάλογο μεταξύ του ΕΚΑ και των, ε, των οργανισμών από το κοινό που μπορεί να μας βοηθήσουν. Οι φιλοδοξίες μας αυτές Επίση, απηχούνται στο πρόγραμμα εργασία μα. Θα ήθελα να σταθώ σε τέσσερα σημεία. Πρώτα απ' όλα, τον, ε, διεθνή αντίκτυπο, τον παγκόσμιο αντίκτυπο του ΡΙΤΣ και του στόχου για το 2020, του τέσσερι στρατηγικού στόχου του ΕΚΑ για τα βιοκτώνα και τι ουσίε PIC, καθώ και την ισορροπία μεταξύ ε, δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω ότι έχει βοηθήσει στο να δημιουργηθούν βασικές αρχές μέσω του ΡΙΤΣ για όλο τον κόσμο και αυτό φάνηκε και από τη συνάντηση SAISM στο Ναϊρόμπι το Σεπτέμβριο. Ήδη πολλοί ε, συντάσσουν τους νόμους τους βασιζόμενοι στις αρχές του ΡΙΤΣ. Εμείς συνεχίζουμε να ασκούμε πίεση και να τους παροτρύνουμε να εφαρμόζουν νόμους που προσωμιάζουν στο ΡΙΤΣ. Αυτό είναι σημαντικό για την ανθρώπινη υγεία ε, παγκοσμίω, για το κοινό μας περιβάλλον, για την αντικονιστικότητα των εταιριών μας και για την καινοτομία εφόσον μπορέσουμε σταδιακά να εξαλείψουμε τις επικίνδυνες χημικές ουσίες. Η συμβολή του ΡΙΤΣ και του οργανισμού μου για τους στόχους του 2020 νομίζω ότι θα μας κάνουν όλους υπερήφανους. Είναι μεγάλη μα χαρά να συνεργαζόμαστε με την ΟΤΟΠΗ και τα κάτι μελη προκειμένου να υπάρχει ένα οδικό χάρτη για το 2020 και να εντοπίσουμε τι χημικέ ουσίε που μα ανησυχούν αλλά και τα σχετικά προβλήματα που προκύπτουν. Ω προ τη βελτίωση υλοποίηση του ΡΙΤΣ, πραγματικά περιμένουμε την αναθεώρηση τη ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ανυπομονησία, διότι έχουμε ήδη, ε, ε, αισθανόμαστε ενθάρρυνση από τι ε, πρώτε εκθέσει, τα πρώτα στάδια που εφαρμογή του ΡΙΤΣ για την ασφαλή χρήση των χημικών ουσιών. Θα πρέπει να προταθούν τρόποι για τη βελτίωση εφαρμογή και υλοποίηση του ΡΙΤΣ. Και αυτό το καλωσορίζουμε. Όμω ε, οι πρόσθετε αιτήσει θα πρέπει να συνοδευτούν και από εγγυήσει για απαραίτητου πόρου. Η στατική μα στόχη τώρα στο πρόσφατο πολιετές πρόγραμμα εργασία μας 2013-2015 και το ετήσιο πρόγραμμα για το 2013 θα δείτε να πηχούνται οι φιλόδοξοι στόχοι. Το πολιετές πρόγραμμα καλύπτει 5 έτη από το 2014 έως το 2018 και διαρθρώνεται γύρω από 4 νέους στρατηγικούς στόχους. Αυτά απηχούν την εμπειρία που έχουμε αποκομίσει ως τώρα με το ΡΙΤΣ και τη συμβολή που είχαμε εμείς ως οργανισμός προκειμένου να πετύχει το ΡΙΤΣ. Όπω θα είδατε από τι γενικέ εκθέσει και τι εκθέσει αξιολόγηση από πέρσι, η πρώτη μα μέρημνα για την επιτυχία του Ρίτς είναι η ποιότητα τη πληροφορία που παρέχεται από πολλέ εταιρείε στα ντοσιέ που τι αφορούν. Η ποιότητα τη πληροφορία είναι πραγματικά θεμελιώ λήθο ε, και έτσι θα δούμε να προκύπτουν ωφέλη από το Ρίτς. Η διαχείριση κινδύνου θα πρέπει να υλοποιείται από τι εταιρείε, ώστε και εμεί να μπορέσουμε να έχουμε ασφαλή χρήση όλων των πληροφοριών στον εργασιακό χώρο. Οι Ευρωπαίοι πολίτε θα πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη ότι τα προϊόντα που αγοράζουν δεν είναι επικίνδυνα για την υγεία των περιβάλλων. Τέσσερι στρατηγικοί στόχοι λοιπόν, ε, συμμόρφωση και ποιότητα στοιχείων για τις, για ουσίες, η αντιμετώπιση της χρήσης των δεδομένων για τις ε, ανισχυτικές, και τις επικίνδυνες χημικές ουσίες, οι επιστημονικές προκλήσεις για τα τοξικά μείγματα και την ε, χρήση ουσιών ε, σε νανομορφές καθώς και αποτελεσματικότητα της εργασίας μας. Όπως σας είπα, πέρσι ασχοληθήκαμε με τα βιοκτώνα και τον κανονισμό και το PIC και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βελτιώσουμε εδώ τις επιδόσεις μας. Όμως πρέπει να σας ε, πω και το εξή εδώ ως προειδοποίηση ότι οι προσδοκίες μας θα πρέπει να είναι σχετικές και με τις δυνατότητες που θα μας δοθούν. Ήδη για το 2013 θα έπρεπε να υπάρχουν περισσότερες θέσεις εργασίας ε, για τα βιοκτώνα. Αλλά υπάρχουν 50, προβλέψεις για 50% μείωση του ε, προσωπικού για το 2013. Ε, και αυτό θα είναι απαραίτητο εφόσον δεν υπάρξουν πρόσθετοι πόροι. Ήδη ένας και μόνο χρόνος για να προετοιμαστούμε για όλο αυτό το εγχείρημα ήταν μια κολοσιαία πρόκληση. Τώρα θα πρέπει να δούμε ότι με τα εργαλεία πληροφορικής οι ε, διαδικασίες που ακολουθήσαμε στο παρελθόν, που δεν ήταν εναρμονισμένες, όπου βασιζόμασταν στη χρήση εγγράφων, έχουν αλλάξει. Θα μπορούσαμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, αλλά εδώ πραγματικά οι επενδύσεις θα πρέπει να είναι ανάλογες των δημοσιονομικών δηλώσεων και θα αργήσουμε να πετύχουμε τους ε, νέους δημοσιονομικούς στόχους. Πάντως ε, τα περισσότερα θα έχουν ήδη ξεκινήσει να υλοποιούνται από το 2013. Θα πρέπει και εσείς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σταθείτε στο θέμα αυτό πολύ άμεσα, γιατί προσφέρουμε βασικές υπηρεσίες και δεν θέλουμε να σας απογοητεύσουμε με το επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρουμε. Ξέρω ότι οι πιέσεις ασκούνται σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν περιμένουμε ιδιαίτερη μεταχείριση ως οργανισμός. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και όρια στο ότι μπορεί να διατεθεί από την πλευρά των πόρων. Όμως η μείωση των κονδυλίων θα πρέπει να ξέρετε ότι θα υποβαθμίσει και τις προσδοκίες που μπορεί να έχει κανείς για την ε, λειτουργία των νομοθεσίας περιχημικών συνολικά. Εξάλλου, δεν είναι ο μόνος τρόπος ε, η εξέβριση περισσότερων πόρων για να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Να σας δώσω ένα παράδειγμα που έχει να κάνει με τον ε, κανονισμό για την φορολόγηση που προκύπτει από τον ΡΙΤΣ. Θα μπορούσαμε εδώ να έχουμε εισόδημα που να προκύπτει και από αυτούς τους φόρους, να τονώσουμε τον ε, θεμητό ανταγωνισμό μεταξύ των εταιριών και να δώσουμε κίνητρα στις εταιρείες να συμμορφώνονται με τις επιταγές μας. Έχουμε εδώ περισσότερες, ε, θα, θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερες εισοδήματα από εταιρείε που δεν αναλαμβάνουν σοβαρά τις ευθύνε τους και οι οποίες μας απασχολούν περισσότερο χρονικά. Ε, όμως έτσι απασχολούν περισσότερο και το δυναμικό και μας απορροφούν περισσότερους πόρους. Ξέρουμε λοιπόν ότι αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει από πολλέ απόψει, εάν επιβάλλονταν φόρε αυτέ τι εταιρείε και από την άποψη του δημόσιου κορβανά και τη ανταγωνιστικότητα και τη δικαιοσύνη βεβαίω. Ω προ τα βιοκτώνα, θα έπρεπε να υπάρχει ένα απλό σύστημα φόρων που να επιτρέπει ένα εύκολο στη διαχείρισή του σύστημα φορολόγηση, ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε το σύστημα που προβλέπεται για το 2013-2014 κατά την υιοθέτηση των κανονισμών για τα βιοκτώνα και που ήδη προβλέπει κάποιες ελάχιστες απαιτήσεις. Προτού αφήσουμε το θέμα των πόρων, να πω ότι το να μπουν οι προπολογισμοί όλων των οργανισμών σε ένα και μόνο σύστημα κοινό είναι κάτι που μπορεί να μην δώσει καλά αποτελέσματα. Είναι κάπως απλουστευτικό, διότι αυξάνονται διαρκώς οι ρυθμιστικές τους αρμοδιότητες. Αυτή η φιλοσοφία του κοινού προπολογισμού ε, ουσιαστικά θα οδηγήσει εσάς και την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο να σταματήσετε να ζητάτε τη δημιουργία νέων οργανισμών με νέες ε, αρμοδιότητες. Θα μπορούσαν όμως να καταρτήσουν αρνητικές προτεραιότητες προκειμένου να υπάρξει εξοικονόμηση πόρων. Η βασική μου ανησυχία για τον ΕΚΑ για την περίοδο 2014-2020 είναι ότι θα υπάρξει μείωση του προσωπικού κατά 5% βάσει πρόταση της Επιτροπής και πάνω από 10% βάσει της πρόταση του Συμβουλίου. Λόγω του ρυθμιστικού του ρόλου θα πρέπει να σκεφτείτε και τις νομικές υποχρεώσεις όμω που έχει αναλάβει ο ΕΚΑ. Και οι γενικέ διευθύνσει, η Γενική Διευθύνση Επιχειρήσεων και Περιβάλλοντο ε, που είναι υπεύθυνε για να μα παρακολουθούν, ξέρουν ότι θα υπάρξουν συνέπειε στην λειτουργία του ΕΚΑ. Είμαστε από τους οργανισμούς που ε, μέσω του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου θέλουμε να πετύχουμε τους ε, φιλόδοξους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει λοιπόν όταν κάνετε αυτές τις δύσκολε επιλογές για την κατανάμε των πόρων να τα γνωρίζετε όλα αυτά και εσεί και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τώρα κάποια σημαντικά στοιχεία από τα περασμένα χρόνια και το, τους φιλόδοξους στόχους μας για τον μέλλον. Κατά πρώτον, ε, πού θέλουμε εσείς να μας βοηθήσετε. Παρακαλούμε να επηρεάζετε όσο μπορείτε σε εθνικό επίπεδο τους υπευθύνου των χωρών σας. Ε, γιατί είναι σημαντικό να έχουμε σχέσεις εταιρικές για την ε, νομοθεσία περί χημικών ουσιών και να υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ εθνικών και ευρωπαϊκών φορέων. Εδώ καταλαβαίνουμε ότι η κατάσταση που αντιμετωπίζουν πολλά κράτη-μέλη είναι δυσχερής επειδή δεν υπάρχουν επαρκείς πόροι σε εθνικό επίπεδο. Οι κανονισμοί δεν ε, υλοποιούνται επιτυχώς. Γι' αυτό σας ενθαρρύνω να ασκήσετε την επιρροή σας ακριβώς της χώρες σας, ώστε η εμπειρογνωμοσύνη μας για τις χημικές ουσίες να διαφυλάσσεται σε κάθε κάτω μέλος. Κατά δεύτερον, σας παροτρύνω και πάλι να μας βοηθήσετε να ευαισθητοποιήσουμε τις εταιρείε τις εκλογικές σας περιφέρειες, να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους και να ασκούν τα δικαιώματά τους, ιδίως τις μικρότερες, αλλά και τους τελικούς χρήστες. Αυτές οι εταιρείε μπορούν να βρουν πληροφορίες σε 23 γλώσσες στον ιστοτοπό μα και να ζητήσουν συνδρομή από τα γραφεία βοήθειας σε εθνικό επίπεδο στη δική τους γλώσσα. Το Κοινοβούλιο, ε, που υπήρξε πάντοτε σταθερός υποστηρικτής του ΡΙΤΣ, Γνωρίζω ότι έχουμε το πλέον εξεχρονισμένο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις χημικέ ουσίες παγκοσμίω. Γι' αυτό λοιπόν είναι κρίσιμη η βοήθειά σας και η φιλία σας. Κάνετε ό,τι μπορείτε, μπορείτε για να βοηθήσετε να φτάσουν οι φιλοδοξίε μα να, να επιτευχθούν. Εδώ θα πρέπει να σκεφτούμε ότι για να έχουμε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες χρειαζόμαστε και ανθρώπινους πόρους και οικονομικούς. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ για την επισκόπηση που μας προσφέρατε. Συζητήσαμε χθες στην Επιτροπή μας για το πώς πρέπει να εφαρμόζεται η νομοθεσία και πώς εφαρμόζεται. Ο οργανισμός χημικών είναι εκ των πυρήνων για την εφαρμογή της νομοθεσίας που έχει εγκρίνει το Κοινοβούλιο. Μιλήσατε για τη χρηματοδότηση βεβαίως πριν από λίγο. Ο οργανισμός σας έχει ανάγκη από την ε, τεχνολογία πληροφορικής για να μπορέσει να λειτουργήσει. Μιλήσατε και για τον προϋπολογισμό και το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Τα καθήκοντά σας έχουμε και μια αξιολόγηση στην ημερήσια διάταξή μας, διότι του χρόνου είναι η πενταετής επέτειος της έγκρισης της οδηγίας REACH από το Κοινοβουλίο. Στην εφαρμογή βεβαίως σημειώνονται προβλήματα υπάρχουν και απώλειες λογοτριβών. Θα δώσω το λόγο τώρα στην κυρία Σάτου Χάση. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Λάνσετ που ήλθε στην Επιτροπή μας για να συνομιλήσει μαζί μας. Είναι σαφές ότι το έργο που επιτελεί ο Οργανισμός Χημικών Είναι κάτι που δεν έχει κάνει καμία χώρα ή καμία περιφέρεια. Είναι σαφές ότι είναι όχι μόνο σημαντικό για μας τους Ευρωπαίους, αλλά και για τον υπόλοιπο κόσμο. Και να γίνει το έργο αυτό σωστά. Και βεβαίως να διδαχθούμε κιόλας από την εμπειρία αυτή. Όπως είπατε και εσείς ο ίδιος, υπάρχουν και σημαντικές ανησυχίες. Μιλήσατε για την ποιότητα των δεδομένων που σας υποβάλλει η βιομηχανία. Θέμα το οποίο έχουμε συζητήσει κατ' επανάληψη και στην Επιτροπή μας και στην διάρκεια επισκέψεων στον Οργανισμό Χημικών. Το θέμα αυτό το περιλαμβάνει και στην επιστολή του ο πρόεδρός μας κύριος Γκρότε που απέστειλε δηλαδή νωρίτερα φέτος. Φαίνεται ότι υπάρχουν πολλές διαστρωματώσεις σε αυτό το πρόβλημα των, ε, της ποιότητας των δεδομένων. Φαίνεται ότι ακόμα και η πληρότητα των δεδομένων που χορηγεί η βιομηχανία δεν ανταποκρίνεται στις νομικές απαιτήσεις. Δηλαδή δεν περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που απαιτούν οι οικίε διατάξεις του κανονισμού REACH. Αυτή είναι η κατάσταση των δεδομένων που έχουμε τώρα από, τον, από τις πρώτες καταχωρήσεις. Θα ήθελα να ακούσω πώς σχεδιάζετε να βελτιώσετε την ποιότητα αυτή στο επόμενο κύμα των καταχωρήσεων που είπατε ότι θα είναι το επόμενο Ιούνιο, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι οι βιομηχανίες δίνουν όλα τα απαραίτητα ε, πληροφοριακά στοιχεία που απαιτεί ο κανονισμός REACH. Το δεύτερο στρώμα, η δεύτερη πτυχή αυτού του προβληματισμού είναι ότι μέχρι τώρα οι επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες έχουν δώσει ατελή έχουν υποβάλει ατελείς φακέλους, μη πλήρης, έχουν υποβάλει φακέλους οι οποίοι όπως εξήγησα δεν είναι δεν πληρούν δηλαδή τα κριτήρια πληρότητος αλλά και ποιότητος. Για παράδειγμα, για περιλαμβάνουν ανεπαρκή μέτρα διαχείρισης του κινδύνου ποιες δράσεις λήφθηκαν, αναλήφθηκαν από τον οργανισμό σας. Έστειλε, στείλατε επιστολές που επισημαίνουν το θέμα και τους επιβάλλουν αυστηρότερα μέτρα τήρησης και διενέργειας των ελέγχων. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι απαραίτητα επαρκές. Εξάλλου, είναι σημαντικό για να είμαστε και δίκαιοι απέναντι στις άλλες επιχειρήσεις οι οποίες υποβάλλουν πλήρης φακέλους. Τι σκέπτεστε λοιπόν να κάνετε, τι σχεδιάζετε να κάνετε για να βελτιώσετε αυτή την κατάσταση. Θα ήθελα επίσης να θέσω και ένα άλλο θέμα εκτός από αυτό το θέμα του προβλήματος δηλαδή της ποιότητας αναφέρομαι στους περιορισμούς ε, για τα χημικά τα οποία είναι γνωστό ότι προκαλούν προβλήματα. Οι πληροφορίες που έχω λέγουν ότι στα έξι χρόνια που ε, είναι λειτουργικός ο REACH, μόνο τέσσερις αποφάσεις έχουν ληφθεί που επιβάλλουν περιορισμούς. Αυτό εμένα μου φαίνεται ότι είναι ε, προϊόν μεγάλης υπερβολικής καθυστέρησης. Ποιος είναι ο λόγος αυτής της αργής πορείας. Είναι επειδή είναι τόσο δύσκολος ο Ρίτς ή επειδή οι επιτροπές της, του ΕΚΑ απαιτούν πολύ υψηλό επίπεδο αποδείξεων πριν να αναλάβουν δράση ή μήπως οφείλεται σε έλλειψη πολιτικής θέλησης από πλευράς ε, χώρων μελών ή και κομισιών. Ευχαριστώ. Κύριο Ζέμπερ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και τον Γενικό Διευθυντή που ήλθε εδώ να συζητήσουμε για τον κανονισμό REACH που νομίζω ότι είναι από τα μεγάλα νομοθετήματα που ενέκρινε η προηγούμενη θητεία. Έχετε και τις πρώτες εμπειρίες. Θα ήθελα να μάθω, κύριε Γενική Διευθυντά, τι γίνεται με την υποκατάσταση που ήταν ένα από τα μέγα θέματα, τα πιο σημαντικές δηλαδή ουσίες, να αντικατασταθούν από άλλες. πώς υποστηρίζει η ΕΚΑ τις επιχειρήσεις οι οποίες κάνουν, προβαίνουν σε αυτή την υποκατάσταση άλλων ουσιών για αυτές που είναι επικίνδυνες. Γιατί ο απότερος στόχος είναι ακριβώς αυτός, να μπορέσουν να εγκαταληφθούν οι επικίνδυνες ουσίες. Ένα δεύτερο, συμφωνώ με την κυρία Χάση, σε ό,τι αφορά τα δεδομένα. Πώς θα διασφαλίσετε ότι η διαχείριση κινδύνου στην οποία προβαίνουν οι επιχειρήσεις θα διευρυνθεί έτσι ώστε και άλλοι ενδιαφερόμενοι να έχουν πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα. Πώς μπορεί να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται ο δημόσιος έλεγχος. Ένα τρίτο θέμα. Χθες ακούσαμε και εγκρίναμε την έκθεση όπου εγώ ήμουν εισηγητής και μάλιστα με μεγάλη πλειοψηφία για την έγκριση ορισμένων ουσιών, με ένα από τα κύρια αιτήματα αυτές τις ε, διασυνδέσεις, αυτά τα cross-links, δηλαδή όταν μια ουσία περιλαμβάνεται στη λίστα προτεραιότητας, που σημαίνει ότι έχει λάβει καταρχήν την έγκριση από τον οργανισμό ΕΚΑ και ενδεχομένως και καταχώρηση, έχει νόημα βέβαια τα δεδομένα αυτά να τα λαμβάνετε και εσείς υπόψη, δηλαδή να έρχονται και σε εσά. Μιλώ για ουσίες στο νερό που προκαλούν προβλήματα, χωρίς να έχουν περάσει από τη διαδικασία αυτή. Τα δεδομένα δηλαδή που συλλέγουν οι επιχειρήσεις διαχείρισης των νερών στις χώρες μέλη, να επανέλθουν στον ΕΚΑ. Πρόκειται για νέο τομέα βέβαια, δεν καλύπτεται από την ισχύουσα νομοθεσία, αλλά μπορείτε ίσως να μας δώσετε μια πρώτη αντίδραση σε αυτή την ιδέα μας, διότι νομίζω ότι είναι σκόπιμο να καταπολεμηθεί η ρήπανση στην πηγή της, στη ρίζα της και όχι στο τέλος, διότι βεβαίως είναι και πολύ πιο οικονομική ε, η αντιρρήπανση στην αρχή. Ευχαριστώ κύριε Ζέμπερ. Στο μεταξύ έχουν έλθει ορισμένοι ε, επισκέπτες από το Πανεπιστήμιο Λέου Βάρντεν, φοιτητές, καλώς ήρθατε, και έχουν προσκληθεί από το συνάδελφο Μπάς Άιχαρτ. Έχουμε επίσης ε, ασκουμένους από τη Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ. Ήρθατε εδώ να δείτε πώς λειτουργεί ο νομοθέτης. Καλώς ήρθατε και εσείς. Και επίσης από τη Γενική Διεύθυνση Διερμηνίας έχουμε επίσης εδώ ε, πρόσωπα τα οποία είναι ασκούμενα. καλώ ήρθατε κι εσείς. Ο Γιώ Λάινεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ντάνσετ, καλώ ήρθατε. Ο ΕΚΑ είναι βασικός οργανισμός για την προστασία του περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι έχουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να διατηρηθεί η αποτελεσματικότητα του οργανισμού σας εκφράσατε τις ανησυχίες σας σχετικά με τη μελλοντική σας χρηματοδότηση και για τα νέα καθήκοντα που ε, συνεπάγεται ο κανονισμός για τα, βιοκτά, τα βιοκτώνα χρειάζεστε βέβαια χρήματα για να δημιουργήσετε ένα μηχανισμό τον οποίο ακόμα δεν διαθέτετε. Εδώ λοιπόν ε, χτυπούν οι κόδωνες του κινδύνου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διότι εφόσον δεν γίνουν αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να υποστηριχθεί η λειτουργικότητα του ΕΚΑ. Μέχρι τώρα ο ΕΚΑ ή και άλλοι οργανισμοί είχε προσόδους και δεν κόστιζε χρήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φαίνεται πως τώρα αλλάζει αυτό τα επόμενα χρόνια και με, με τον κανονισμό και τα λοιπά και πρέπει να φροντίσουμε η χρηματοδότηση να είναι επαρκής ώστε να μην περικόπτει τις δραστηριότητέ σας. Είπατε κι εσείς ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει ρόλο πρωτοπόρο παγκόσμια για την ρύθμιση των σχετικών με τις ε, χημικές ουσίες. Τι κάνουν άλλες περιοχές του κόσμου. Παλαιότερα ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες η ηγέτητα δύναμη σε ζητήματα ρύθμισης των χημικών. Τώρα γίνονται και εκεί ορισμένα πράγματα, καθώς και στην Κίνα. Το ερώτημα είναι τα χημικά τα οποία εμείς απαγορεύουμε, αλλά επιτρέπουν τη χρήση τους. Άλλοι ενδέχεται με, μέσω εισαγόμενων προϊόντων να επανέλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς λοιπόν θα εμποδίσουμε εμεί με να κάνουμε το καλό, άλλοι όμω οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται τελικώ να μα δηλητηριάζουν. Θυμίζω τα παιδικά παιχνίδια, τα εφάσματα και άλλα σχετικά παραδείγματα. Επίση, αναφέρθηκε προηγούμενα συνάδελφό μου στην υποκατάστατη, στην υποκατάσταση, συγγνώμη. Είπατε κι εσεί ότι θέλουμε ασφαλέστερα χημικά. Άρα, ορισμένα πρέπει να εξαφανιστούν από τα ράφια και να αντικατασταθούν από άλλα. Αναρωτιέμαι και εγώ γιατί κινείται τόσο αργά αυτή η υποκατάσταση. Επίσης, πιο επίκαιρο ερώτημα για την χρήση χημικών στον θρηματισμό, στο fracking των σχιστολίθων δηλαδή. Εκεί υπάρχει η ανησυχία ότι χρησιμοποιούνται χημικές ουσίες οι οποίες ενδεχομένως είναι προβληματικές. Και δεύτερον, δεν είναι γνωστό το τι μπορεί να προκαλέσουν. Τι νομίζετε. Ευχαριστώ. Κράμερ. Ευχαριστώ. Πρώτα εκφράζω τον ε, σεβασμό μου για, τα, για το έργο σας, διότι έχετε αναλάβει ένα πραγματικά τεράστιο καθήκον. Δεύτερο, σε όλη την θητεία σας ως διευθυντού του ΕΚΑ έχετε λάβει πάντοτε πολύ σοβαρά υπόψη το Κοινοβούλιο. Πάντοτε φροντίσατε ώστε και να ζητάτε τη συμπαράστασή μας και να αποδίδετε και λογαριασμό στο Κοινοβούλιο. Κάτι το οποίο σας διακρίνει βεβαίως από άλλους διευθυντές οργανισμών. Συγκεκριμένο ερώτημα τώρα για την λίστα του παραδείγματος 14, στην οποία αναφερθήκατε και εσείς στην ομιλία σας. Όλο και περισσότερο μας προσεγγίζουν επιχειρήσεις που εκφράζουν ανησυχίες ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν απαγορεύσεις υλών για τις οποίες δεν έχουν εναλλακτικές επιλογές. Ένα επίκαιρο παράδειγμα που έφτασε στο γραφείο μου είναι ενώσεων του χρωμίου και του στρόντσιουμ χωρίς να πω σε λεπτομέρειες, ωστόσο ενδέχεται εδώ να έχουμε μια παράπλευρη ζημιά, η οποία δηλαδή ούτε το περιβάλλον εξυπηρετεί, ούτε τη βιομηχανία. Χρησιμοποιούνται τέτοιε ουσίε, για παράδειγμα, για την συντήρηση των αεροσκαφών ω αντιοξυδοτικά. Και ενδέχεται να υπάρξει ο κίνδυνο η συντήρηση των αεροσκαφών να βγει από το πεδίο εφαρμογή του ΡΙΤΣ. Δεν ξέρω αν μπορείτε να απαντήσετε βέβαια τώρα. Αλλά διερωτώ με πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που αναφέρονται στην λίστα αυτή που συμπεριλαμβάνει τις διάφορες ύλε. Λαμβάνονται πάντα υπόψη όλα τα υπέρ και τα κατά, οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι για το περιβάλλον αλλά και για την οικονομία κλπ. Διότι εν τέλει ποιο θα είναι το όφελο για την Ευρώπη αν στο μέλλον η συντήρηση των αεροσκαφών γίνεται, γίνεται για παράδειγμα στην Τουρκία. Και έτσι εκεί υπάρχει επιβάρυνση του περιβάλλοντο, ενώ εμεί εδώ απαγορεύουμε τη χρήση των ουσιών αυτών. Δεν νομίζω ότι ωφελεί κιόλα τις επιχειρήσεις να περιμένουν την διαδικασία έγκρισης και στο μεταξύ σχετικέ επενδύσει για τι εγκαταστάσει που είναι απαραίτητε για τη συντήρηση αεροσκαφών, στο παράδειγμα αυτό, να γίνουν εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Έχω πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις και δεν συνδέονται άμεσα με τις δραστηριότητες της, του οργανισμού σας, αλλά με την πιθανή μόλυνση ε, από χημικά. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο θαύτηκαν πολλά χημικά όπλα στην περιοχή μας, στη Βαλτική. Και τώρα ένα τμήμα του αγωγού του Nord Stream έχει τελειώσει και ένα άλλο ε, φτιάχνεται στην περιοχή του Καλίνιγκρατ. ε, φτιάχνοντας αυτόν τον αγωγό μπορεί να αγγίξουμε τις αποθήκες που έχουν θαυτεί, αποθήκες που έχουν θαυτεί αυτά τα χημικά όπλα. Και επομένως ε, μπορεί να υπάρξει χημική μόλυνση. Ο οργανισμός σας έχει εμπειρία από την επίλυση τέτοιων προβλημάτων. Έχει συμβεί κάτι αντίστοιχο στο παρελθόν ποτέ. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω δεν είσαστε πολύ δραστήριοι στην διάλυση χημικών όπλων, αλλά η χημική μόλυνση είναι τμήμα της εντολής σας, των αρμοδιοτήτων σας. Ε, ζητώ συγγνώμη που πρέπει να φύγω τώρα, θα πρέπει να πάω να ψηφίσω. Απαντήστε όμως αυτή την ερώτηση, γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θέλουν να ακούσουν την απάντηση και θα μου το διαβιβάσουν. Συναντηθήκαμε και νωρίτερα και έκανα τις, ε, και τις ερωτήσεις μου προηγουμένως. Ξέρετε για αυτή την έκθεση μια μη κυβερνητική ε, οργάνωση, ξέρετε για τη σύγκρουση συμφερόντων και τι κάνετε εσεί προληπτικά και πώς ε, μεταφέρουμε ε, χημικές ουσίες από τον ε, κατάλογο ας πούμε και, τα, και υποβάλλουμε αυτές τις ουσίες σε περισσότερους περιορισμούς. Ε, πόσες ουσίες έχουμε σε αυτόν τον κατάλογο, προσωρινό κατάλογο του 2015 ehemaligen äh, Ευχαριστώ. Ποιος θέλει να πάρει το λόγο? Ο κύριος Σιμάνσκι. Συμφωνώ απόλυτα με την παρατήρηση που έγινε για τη Βαλτική θάλασσα. Υπάρχει ένα πραγματικό πρόβλημα, ένα κολοσιαίο πρόβλημα και αυτό γίνεται ακόμα μεγαλύτερο γιατί δεν ξέρουμε ακόμα ποια είναι η ποσότητα των επικίνδυνων αποβλήτων που έχουν χυθεί στις, ε, στη Βαλτική θάλασσα. Δεν ξέρουμε τι έχουν κάνει οι Ρώσοι, αλλά υπάρχουν, υπάρχει και η διάβρωση, η οποία δημιουργεί πρόβλημα σύν χρόνο. Δεν ξέρουμε ποιος έχει ρίξει τι, πόσο έχει ρίξει. Μην, ξε, μην ε, ξεχνάτε ότι η Βαλτική είναι μια θάλασσα κλειστή ουσιαστικά. Υπάρχουν δύο περιοχές που χωρίζουν τη Βόρεια Θάλασσα από την ε, Βαλτική. Ε, εκεί περνάει πολύ λίγο νερό και μπορεί να δημιουργηθούν τεράστιες ε, περιβαλλοντικές καταστροφές. Είχαμε περιπτώσεις στην Πολωνία όπου ψαράδες κάηκαν από προϊόντα που βρισκόταν μέσα στη θάλασσα θα πρέπει να εγγύψουμε σε αυτό το πρόβλημα που είναι πολύ σημαντικό, που έχει τεράστιο κόστος και που απαιτεί συνεργασία αλλά και κουράγιο. Πολύ συχνά όταν ε, ρίχνουμε ουσίες στη θάλασσα δεν παίρνουμε καμία ευθύνη. Αυτό το κάνανε πολύ τα κομμουνιστικά καθεστώτα. Αλλά θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα να δράσει για να βοηθήσει τις χώρες της Βαλτικής. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι το εξή μετά από αυτά που είπε η συνάδελφος. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα. Έχετε προβλέψει δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση γιατί μπορεί να πρόκειται για μια ορολογιακή βόμβα εδώ στη Βαλτική. Ότι θα πρέπει να διευρυνθεί η εντολή της ΕΚΑ ώστε να προβαίνει και στην εκαθάριση πολεμικών υλών. Τώρα, εκπρόσωπός μας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ήταν και παλαιότερα Ευρωβουλευτής, η κυρία Αν και βεβαίως είναι ε, καλά γνωστή σε όλες και όλους μας. Ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Να... ήρθαμε μεγάλη χαρά εδώ, ε, ακόμα μεγαλύτερη είναι αυτή η χαρά γιατί βλέπω και πολλούς γνωστούς εδώ και βλέπω ότι η Επιτροπή σας δουλεύει εργοδός για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος. Θέλω να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε την εντολή να συμμετάσχω στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΑ. Εγώ ανέβηκα καθοδόν ε, μετά την συναδέλφο Κριστίνα Ρούντεν και εντυπωσιαστήκαμε από τη δουλειά που κάνει ο οργανισμός υπό την διεύθυνση του Γκέρτ ε, Ντάντσερτ. Έχουμε 30.000 ουσίες, 600 άτομα, έχουμε ένα σύστημα πληροφορικής περίπλοκο. Νομίζω ότι πρέπει τουλάχιστον να χαιρετήσουμε τη δουλειά που κάνει ο οργανισμός. Θέλω να στηρίξω αυτά που είπε ο διευθυντής μας. Υπάρχει ένα θέμα οικονομικό, χρηματικό. Και παρά τις περικοπές που ζητάμε ε, και στα κράτη-μέλη και στη δημόσια διοίκηση, πρέπει να κάνουμε προσπάθεια, αν θέλουμε, ε, να ασχοληθούμε με τον έλεγχο των διοκτώνων και των νανοηλικών και γι αυτό, για να γίνει αυτό θα πρέπει να δώσουμε τα απαραίτητα χρήματα στον οργανισμό. Όταν ε, επισκέφθηκε η αντιπροσωπή σας τέλος Αυγούστου την υπηρεσία, Τέθηκαν κάποιες ερωτήσεις, η κυρία Σάτο να έκανε την ερώτηση, είναι το compliance check, ο έλεγχος συμμόρφωσης. Επαναλαμβάνω ότι εγώ δεν ξεκίνησα από την αρχή στον ΕΚΑ. Πρέπει να δούμε αυτό το θέμα σε επίπεδο νομοθεσία. Ζητάμε από τον οργανισμό να ελέγξει το 5% των φακέλων. Ο, η ποιότητα των φακέλων επαληθεύεται από τις αρχές των κρατών μελών, αν κατάλαβα καλά. Σήμερα τα πράγματα είναι πολύ περίπλοκα, γιατί ε, υπάρχουν φάκελοι ατελεί. Ο έλεγχος ε, δεν γίνεται με γραμμικό τρόπο. Ε, ε ελέγχουμε και την ε, γραπτή δήλωση. Συχνά έχουμε χιλιάδες φακέλους και δεν μπορούμε να ελέγξουμε μόνο μέσω της πληροφορικής τα πάντα. Αν θέλουμε να κάνουμε πραγματικά ποιοτικό έλεγχο συμμόρφωσης στο 100% των φακέλων, θα πρέπει, νομίζω, να δημιουργήσουμε ένα σύστημα πληροφορικής πολύ επαχθές για να ε, επαληθεύουμε κάθε τραγωνίδιο. Αυτό απασχολεί και το Κοινοβούλιο και τον Οργανισμό και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Υπάρχει μια ομάδα εργασίας που ασχολείται με το θέμα αυτό για να καταλάβουν τις δυσκολίες των επιχειρήσεων για να συμπληρώσουν σωστά τους φακέλους από την πρώτη φορά και να εμποδίσουμε τον οργανισμό να ε, τις καταγγέλει και να βλέπουμε, εν πάση ποιες είναι οι επιπτώσεις. Σημαντικό αυτό. Εμείς παρεμβαίνουμε και δρούμε ανεξάρτητα, παρότι επηρεαζόμαστε προφανώ ο καθένα από το παρελθόν, το εγώ από τα πέντε χρόνια που πέρασα στο Κοινοβούλιο, Πρέπει να πω ότι υπάρχουν κάποιε ανησυχίε ε, από πλευρά βιομηχανία, κυρίω για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Έχουμε δημιουργήσει δηλαδή ένα πολύ περίπλοκο σύστημα, πλήρε, και για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει φανταστείτε το εξή, ότι οι εκθέσει για την ε, χημική ασφάλεια ή τα δελτία δεδομένων ε, που αφορούν την ασφάλεια των προϊόντων είναι φάκελοι πολύ δύσκολοι, πολύ περίπλοκοι, που φτάνουν και τις 300 σελίδες. Φανταστείτε λοιπόν τι σύστημα δημιουργήσαμε. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να χαιρετήσουμε τη δουλειά που έγινε, το σύστημα της πληροφορικής που, χρησιμοποιείται και τη δουλειά του οργανισμού και του προσωπικού που έχει σαν στόχο και πρέπει να το επαναλάβουμε, να γίνει ε, οργανισμός διεθνής για τα χημικά προϊόντα. Και θα πρέπει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να μην το ξεχνάνε αυτό. Αν θέλουμε να κρατήσουμε τη βιομηχανία μας, αν θέλουμε να διατηρήσουμε την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, θα πρέπει η Ευρώπη να παίξει πρωταρχικό και ηγετικό ρόλο. Γι' αυτό λοιπόν ε, σας καλώ να στηρίξετε αυτόν τον στόχο του οργανισμού. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βίλμουντ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν έχω να, πάω, να πω πολλά πράγματα, να αντιδράσω στα σχόλια για τους πόρους, που φυσικά είναι αρμοδιότητα της Κομισιόν. Για τα βιοκτώνα, δεν είναι κανένα από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος για να σας δώσει πληροφορίες για την κατάσταση των βιοκτώνων για τον κανονισμό για τα τέλη, τον κανονισμό REACH, στον οποίο αναφέρθηκε ο Διευθυντή. Είχαμε κάποιες χρήσιμε ανταλλαγέ απόψε με την ΕΚΑ για το πώς θα μπορούσαμε να αναθεωρήσουμε αυτόν τον κανονισμό για τα τέλη. Καταλαβαίνουμε την επιθυμία του ΕΚΑ να μεγιστοποιήσει του πόρου του, αλλά πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στις απαιτήσει του κλάδου και στους πόρους του ΕΚΑ και πρέπει να σεβόμαστε και τα νομικά κείμενα που περνάνε από το Κοινοβούλιο και το ε, Συμβούλιο που περιορίζουν την ελευθερία μας. Για τις εκτόσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε ο κ. Ντάνσερ. Δεν χρειάζεται να σας πάρω περισσότερο χρόνο, γιατί νομίζω ότι ο Διευθυντής μπορεί να σας απαντήσει. Αν οπωσδήποτε όμως θέλετε τη βοήθειά μου, μπορώ να ξαναπάρω το λόγο. Ευχαριστώ και εγώ, λέει ο Πρόεδρος, ο κύριος Ντάνσετ. Um, Ευχαριστώ. Να ξεκινήσω πρώτα απ' όλα με τις ερωτήσεις που μου τέθηκαν. Πρώτα απ' όλα ερωτήσεις της κυρίας Χάσιο. Ανησυχήσατε για τους ελέγχους πληρότητας, μετά τους ελέγχους συμμόρφωσης και μετά για την ποιότητα των πληροφοριών σε σχέση με τα θέματα αυτά. Ως προς την πληρότητα, συζητήσαμε επανειλημμένως με τους ενδιαφερομένους και το Διοικητικό Συμβούλιο για το τι εννοούμε με την πληρότητα και αν συμμόρφωση αποτελεί πληρότητα και καταλήξαμε ότι η πληρότητα είναι να δούμε αν παρέχονται όλα τα τμήματα ενός φακέλου. Αλλά η συμμόρφωση ελέγχεται με, την, με τους σχετικούς ελέγχους συμμόρφωσης επίσης. Να έχουμε υπόψη ότι η πληρότητα γίνεται με τρόπο αυτοματοποιημένο. Χιλιάδες φάκελοι φτάνουν ταυτόχρονα. Οι εταιρείε πρέπει να μπορούν να προβλέψουν πότε θα είναι πλήρη η θάκελη που αποστέλουν και τι αποτελέσματα να περιμένουν στους ελέγχους πληρότητας. Προσπαθούμε να έχουμε όλο και καλύτερα αποτελέσματα ως προς την πληρότητα και έχουμε και σχέδια για το μέλλον για να βελτιώσουμε τους ελέγχους πληρότητας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε σταδιακά. Βεβαίως, όπως είπα και προηγουμένως, το μορατόριο για την επόμενη προθεσμία καταγραφής ε, αρχίζει από αύριο. Οπότε θα έχουμε νέους ελέγχους πληρότητας σε έξι μήνες. Τώρα για, τα, για τους φακέλους όπου δεν υπάρχει συμμόρφωση. Εδώ μαθαίνουμε και μέσα από τις εμπειρίες μας. Εξετάζουμε όλα τα θέματα σε όλες τους τις πτυχές όλες τις πτυχές των φακελών και έχουμε κάποιες πρώτες ήπιες στάσεις με επιστολές για την ε, παρακολούθηση της ποιότητας. Τώρα σιγά σιγά ε, απομακρυνόμαστε από αυτό και ασχολούμαστε με την έλλειψη ε, συμμόρφωσης. Διότι κατά πρώτον χρειάζονται ορθές πληροφορίες βάσει των σχετικών απαιτήσεων προτού γίνει μια πλήρες αξιολόγηση των οδηγιών ασφάλειας. Γι' αυτό η συμμόρφωση πλέον έχει συγκεκριμένου στόχους. Πρώτα ε, επικεντρωνόμαστε στι απαιτήσει πληροφοριών και μετά στις οδηγίε ασφάλεια. ασφάλειας. Προχωρούμε βήμα-βήμα πάντως και ελπίζουμε ότι θα καλύψουμε όλους τους φακέλους που μπορεί να έχουν ε, προβλήματα. Όμως όταν εντοπίζουμε ντοσιέ που σε γενικές γραμμές ε, παρουσιάζουν καλή συμμόρφωση αλλά έχουν συνολικώ κακή ποιότητα Οπότε έτσι γίνονται μη συμμορφούμενα. Εκεί λαμβάνουμε ήπιες αποφάσεις και απευθυνόμαστε άμεσα σε αυτό. Ή μπορεί να απειλήσουμε και με περαιτέρω δράση εναντίον των εταιριών αυτών. Αλλά αυτά είναι κάποιες δεκάδες ντοσχέ και φανταστείτε πόσο διαφορετικό είναι όταν αντιλαμβάνουμε χιλιάδες ντοσχέ. Είναι πολύ μικρό λοιπόν το τμήμα της μη συμμόρφωσης. Επίσης προσπαθούμε να αφήσουμε τα, σε τις επιστολές για την ποιότητα κατά μέρο και να έχουμε περισσότερο ήπιες αποφάσεις για τους περιορισμούς. Όταν ε, είπαμε ότι το REACH λειτουργεί εδώ και 5 ή 6 χρόνια, τι σημαίνει αυτό. Ότι τον ερχόμενο Ιούνιο θα κλείσουν 5 χρόνια λειτουργίας του REACH και ελπίζω να το γιορτάσουμε εδώ και στο Κοινοβούλιο ως τώρα τέσσερις, νέου, τέσσερις νέους περιορισμούς προτείναμε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία τώρα είναι στη φάση έγκρισης των αποφάσεων αλλά πρέπει να σκεφτεί κανείς το εξή. Ότι υπάρχει εδώ μια συγκεκριμένη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείτε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα προηγούμενα χρόνια είχε εγκρίνει περισσότερους περιορισμούς κατάλοιπο παρελθόντος. Χρειάζεται λοιπόν και χρόνος για την έγκριση των επίσημων αυτών αποφάσεων από την Επιτροπή. Είναι χρονοβόρες οι διαδικασίες αυτές. Ο κύριος Σλίτερ ανέφερε άλλες, άλλους περιορισμούς που προκύπτουν από την νομοθεσία που ίσχυε προηγουμένως. Οι πρώτες τελικές αποφάσεις πάντως είναι πολύ ε, κάτι πολύ πρόσφατο. Πάντως, το πλαίσιο μας είναι πολύ αυστηρό λόγω της νομοθεσίας. Συνεχώς έχουμε να τηρούμε προθεσμίες. Μόλις φτάσει κάτι στα χέρια μας, πρέπει να μπορούμε να προβλέψουμε λίγο πολύ πότε θα είναι έτοιμες οι γνωμοδοτήσεις. Και έπειτα απαιτείται χρόνος για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου εκεί όμως δεν υπάρχει καταλεκτική ημερομηνία για τη λήψη απόφαση μέσω επιτροπολογία. Έπειτα για την υποκατάσταση, Πώ μπορούμε να βοηθήσουμε. βεβαίω και μπορούμε να βοηθήσουμε ενημερώνοντα κατά πρώτον. Ενημερώνοντας τον κατάλογο των υποψήφιων ουσιών, των εγκεκριμένων και δίνοντας κίνητρα στις εταιρείε αρκετά νωρίς ώστε να ξεκινήσουν τις προσπάθειες υποκατάστασης. Πρέπει όμως κανείς να συνειδητοποιήσει ότι το θέμα αυτό έχει ιδιαίτερα τεχνικό χαρακτήρα. Διότι πρέπει να λάβει χώρα εντό των εταιριών σε επίπεδο εταιρεία και δεν πρέπει να υπάρχει και απόρριτο τη ανταλλαγή μια ουσία με μια άλλη. Αυτό ουσιαστικά θα είναι και μια απόδειξη του κατά πόσο είναι ευφυή μια εταιρεία στο να αντιμετωπίσει του ανταγωνιστέ τη εγκαίρω. Επίση πρέπει να τονίσουμε ότι το REACH έχει δώσει φοβερά κίνητρα για την υποκατάσταση ω τώρα. μισές από τις ε, καταχωρημένες ουσίες έχουν ήδη εγγραφεί. Οπότε είναι πολλές εταιρείε που εκμεταλλεύτηκαν τις προθεσμίες που προβλέπει η νομοθεσία ώστε να κινηθούν γρήγορα στην υποκατάσταση. Γρηγορότερα από ό,τι θα φανταζόταν κανείς. Ως προς τις πληροφορίες και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την διαχείριση των κινδύνων. Πρώτα απ' όλα, η διαχείριση του κινδύνου απευθύνεται και στι δημόσιε αρχέ. Γι' αυτό θέλουμε οι δημόσιες αρχές να έχουν πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που διαθέτουμε εμεί. Εκείνοι θα αναλάβουν τι πρωτοβουλίε για τη διαχείριση κινδύνου. Από κοινό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουν πλέον λοιπόν πλήρη πρόσβαση στα συστήματά μα και του διευκολύνουμε και στο πώ μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτέ τι πληροφορίε, Να δουν τι είναι το λογικότερο να κάνουν για να προχωρήσει η διαχείριση αυτή. Μάλιστα τώρα, φέτος μόλις, άρχισαν ε, να κάνουν αξιολόγηση ουσιών τα κρατημέλη. Παίρνουν όλες τις πτυχές μιας ουσίας και εξετάζουν εάν οι πληροφορίες που παρέχονται παρουσιάζουν ελλείψεις. Αναλύουν λοιπόν τους διάφορους ε, φακέλους, τα διάφορα θέματα για να δουν κατά πόσον χρειάζεται περισσότερες πληροφορίες. Είναι πάντως σημαντικό οι φάκελοι καταχώρησης να είναι κανείς ποιότητας. Θέλουμε πληροφορίες υψηλής ποιότητας. Δεν κατάλαβα πολύ καλά το τρίτο σας ερώτημα, αλλά ελπίζω να το καλύψουμε διμερώς. Ήταν αρκετά συγκεκριμένο, οπότε ας το συζητήσουμε μετά τη λήξη της συνεδρίασης ε, διμερώς για τη χρηματοδότηση. Ήδη ανέπτυξε το επιχείρημα για το εξή. Δεν είναι επαρκή η χρηματοδότηση για τα βιοκτώνα, από τη μια. Και έχω εκφράσει τι σοβαρέ μου ανησυχίε και στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντο. Θα δούμε αν θα βρούμε λύσει τι ερχόμενε εβδομάδε. Πάντω, αυτό που χρειάζεται είναι κι εσείς να βεβαιωθείτε ότι ολόκληρο το κονδύλι θα εγκριθεί από το 2013, τουλάχιστον από τη δική σας πλευρά. Οποιαδήποτε περικοπή θα πλήξει ιδιαίτερο την προετοιμασία για την υλοποίηση αυτού του νέου, της νέας, αυτής της νέας νομοθεσίας που αναλαμβάνουμε να εφαρμόσουμε κι εμείς. Επίσης μιλήσατε για τη διεθνή συνιστόσα. Πώ αντιδρούν άλλε χώρε κατά κύριο λόγο οι Ηνωμένε Πολιτείε και Κίνα. Γνωρίζουμε ότι οι χώρε αυτές ήδη προετοιμάζονται για την ενδεχόμενη, για την ευρωπαϊκή νομοθεσία που ενδεχομένως θα τεθεί σε ισχύ. Βεβαίως, η νέα νομοθεσία στι χώρε αυτέ, ε, στι ΗΠΑ λόγω χάρη, άρχισε να εξετάζεται πριν δύο χρόνια. Πρέπει να, να έχουν όμω και κοινοβουλευτική έγκριση. Και πρέπει να δούμε κι εμεί αν όντω θα προχωρήσουν σε αναθεώρηση τη δική του οδηγία. Γιατί και για μα είναι πολύ ενδιαφέρον να έχουν εξυγχρονισμένα νομοθετικά μέτρα ώστε να μπορούμε να έχουμε ανταλλαγή απόρριτων πληροφοριών. Θέλουμε να μπορούμε να έχουμε ανταλλαγή στοιχείων να εκμεταλλευτούμε τον πλούτο που υπάρχει από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να το κάνουμε λοιπόν αυτό και πραγματικά ανυπομονούμε να υπάρξει πρόοδος εδώ. Επίσης η Κίνα με τη νέα ηγεσία τώρα θα δεχτεί πιέσει να έχει λιγότερο προστατευτική και καλύτερη νομοθεσία για την ε, αγορά των χημικών. Τα δούμε. Και η Ινδία προχωρά προς την κατεύθυνση αυτή του ΡΙΤ. Άλλη μεγάλη δύναμη στην ε, μελλοντική αγορά. Οικονομική δύναμη που θα μπορούσε να ωφελήσει εφόσον αναθεωρήσει την νομοθεσία της. Βεβαίως, σημαντικό για μας είναι να μπορούμε να συνεργαστούμε στενά όχι μόνο με τις αρχές που πραγματοποιούν τους ελέγχους στο επίπεδο της παρασκευής ουσιών, αλλά και με τις τολωνιακές αρχές. Γι' αυτό εντείνουμε τη συνεργασία μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε και τελωνιακές διατάξεις να συμβαδίζουν με το τι κάνουν ε, και οι υπόλοιπες αρχές στους άλλους τομείς ελέγχου. Ως προς την υποκατάσταση ελπίζω ότι απήντησα τώρα για το θρηματισμό. Πραγματικά αυτό το σημείο είναι πολύ δυσχερές. Η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος ζήτησε να ασχοληθούμε με το θρηματισμό. Μας ζητήθηκαν πληροφορίες. Εξετάζονται αυτή τη στιγμή τα σχετικά ντοσιά για να δούμε τι πληροφορίες μπορούν να αντιληθούν από αυτά. Όμως μιλάμε για εξαιρετικά λεπτομερή και συστηματική χρήση μιας πολύ συγκεκριμένη ουσίας και δεν υπάρχει από τη στιγμή καμία απέτηση, καμία οδηγία ασφαλείας για κάθε λεπτομερή χρήση μιας συγκεκριμένης ουσίας. Η, ο μηχανικός κλάδος ε, έχει το δικαίωμα να συνοψίζει τις χρήσεις μιας ουσίας. Οπότε πολλές βασικές πληροφορίες μπορεί να χαθούν στο μεταξύ. Γι' αυτό λοιπόν στο μέλλον θέλουμε να μπορούμε να συζητήσουμε με τις εταιρείε χημικών πώς θα έχουμε πιο συγκεκριμένη περιγραφή για να έχουμε και ανάλογες οδηγίες ασφαλείας για τους χρήστες. Αυτό είναι μέρος του ερχόμενου πολιετούς ε, προγράμματος εργασιών. Για το 2014 θα μας απασχολήσουν και παράπονα εταιρεών που παράγουν λόγω χάρη ουσίες χρωμιούχες. που χρησιμοποιούνται σε διάφορες επιφάνειες και πολλές φορές και στην ε, παραγωγή αεροσκαφών. Εδώ είναι υπερβολική αυτή η αντίδραση και έχουμε και πλήρη, παρανόηση του τι γίνεται από την πλευρά της ε, έγκρισης. Η έγκριση, η εξουσιοδότηση σκοπό έχει να δώσει κίνητρα για την υποκατάσταση. Οι εταιρείε δεν πρέπει να το αντιλαμβάνονται αυτό ω πλήρη απαγόρευση, παρόλο που αυτό του συμβαίνει κάποιε φορέ. Όχι, δεν είναι σκοπό η εξουσιοδότηση να χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για την πλήρη απαγόρευση. Την υποκατάσταση θέλουμε να ενισχύσουμε. Ε, ο βιομηχανικός αυτός κλάδος θα πρέπει να διεξάγει τη σχετική έρευνα, ενώ υπάρχει η εξουσιοδότηση και ισχύει. Υπάρχουν απλώς χρονικά όρια και πρέπει να προχωρήσουν στην εξέταση του θέματος μαζί μας μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Νομίζω ότι υπερβάλλουν πάντως. Θα πρέπει να φοβούνται λιγότερο τις ε, εφαρμογές της εξουσιοδότησης. Ναι. Εδώ λοιπόν οι εταιρείε πάντοτε αναζητούν ένα χρονικό πλαίσιο προκειμένου να κάνουν την αποκατάσταση πριν λήξει η προθεσμία για την εξουσιοδότηση. Σπάνια λοιπόν έχουμε αιτήσει πολύ νωρίτερα από ό,τι αρχικά προβλέπαμε. Τώρα σε ό,τι αφορά τη ρήπανση στη Βαλτική και τα όπλα, όπως είπατε και εσείς Πρόεδρε, δεν είμαστε αυτομάτως ε, αρμόδιοι γι' αυτό. Προσπαθούμε να βεβαιωθούμε ότι είναι σωστά τοποθετημένα στον κατάλογο οι ουσίες. Να έχουν βλαπτικέ συνέπειες για το σύστημα, το υδάτινο. Μια αν γίνονται σεβαστέ οι σχετικές οδηγίες για τα ύδατα. Αλλά εκεί περιορίζεται το έργο μας. Ο κύριος Λίτερ επίση. ανέφερε την ε, σημασία της σύγκρουσης ε, συμφερόντων. προσέχουμε ιδιαίτερος ώστε να μην προκύψει σύγκρουση συμφέροντος και γι' αυτό διαχειριζόμαστε πολύ προσεκτικά τη σύνθεση των πάνελ, την συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, συγκρίνουμε τις δηλώσεις συμφερόντων τώρα για τις χημικές ουσίες των κατάλογο των υποψήφιων ουσιών. για μας θα ήταν καλό να περάσουν πολύ γρήγορα, να περνάνε πιο γρήγορα οι ουσίε από τον κατάλογο των υποψήφιων ουσιών στον κατάλογο των ε, εγκεκριμένων. Διότι υπάρχει ο χρόνος για τις, ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο για τη σύσταση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξέρει πολύ καλά ότι υπάρχουν εταιρείε που αντιστέκονται, δεν θέλουν να μπουν στον κατάλογο τη εξουσιοδότηση. Πόσε ουσίε θα έχουμε στο 2015 στον κατάλογο των υποψήφιων ουσιών μέσα στην ερχόμενη τριετία, δύσκολο να μιλήσω με αριθμό εδώ και να, είχα, να έχω ποσοτικού στόχου. Ελπίζω να έχουμε τι σωστέ ουσίε. Αυτέ που πραγματικά ξεχωρίζουν και χρησιμοποιούνται ευρέω και πραγματικά επηρεάζουν την καθημερινή ζωή των πολιτών. Θέλουμε εδώ να στηρίξουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κάτι μέλη με ένα νέο προγραμματισμό που θα εξετάσουμε θέματα και το σχέ όπου γνωρίζουμε ότι αφορούν ουσίες που παρουσιάζουν ε, ιδιαίτερε ιδιαίτερες ανησυχίες. Θα πρέπει λοιπόν τα κράτη-μέλη να αποφασίσουν μετά εάν θα ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο ή το δρόμο της πλήρους απαγόρευσης. Είναι και αυτό ιδιαίτερα σημαντικό. Επίσης, η κυρία στήριξε το έργο μας. Όντως, έχουμε πολλά να κάνουμε, έχουμε μεγάλο φορτό εργασίας, προσπαθούμε να προωθήσουμε όλες αυτές τις, όλα αυτά τα θέματα. Και θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε με φιλοδοξία τους στόχους μας. Τώρα για τους ελέγχους συμμόρφωσης, πραγματικά θα ήταν πολύ λυπηρό εάν στο τέλος προκύψει ευρύτερο πρόβλημα. Με την ποιότητα των ε, θεμάτων, των ντοσιέ και με την συμμόρφωση. Συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να παραμείνει το προσωπικό που ασχολείται με την αξιολόγηση και να κάνει και περισσότερα από ό,τι αρχικά προβλέπεται νομοθετικός. κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να έχουμε μεικτή χρηματοδότηση, δημόσια και ιδιωτική, όπως τονίζω εδώ και πολλή ώρα, και να λειτουργούμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Είπατε ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα ώστε οι εταιρείε να ετοιμάζουν εκθέσει για την ασφάλεια των χημικών ουσιών και τα σχετικά δελτία. Αυτό το προγραμματίζουμε. Όμω σημαντικό είναι και οι εταιρείε να κινούνται γοργά, να αναπτύσσουν τα δικά τους εργαλεία και να ετοιμάζουν τα δελτία για την ασφάλεια των χημικών ουσιών και για άλλους. Υπάρχει τυποποιημένο λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται σε αυτά τα δελτία, οπότε αυτό καλό θα ήταν να το γνωρίζουν ε, οι ενδιαφερόμενες εταιρείε. Εμείς φροντίζουμε να γίνονται γρήγορα μεταφράσεις και η συλλογή των στοιχείων απευθυνόμαστε διαρκώς τις εταιρείες ώστε να συνεχίζουν διαρκώς αυτές τις προσπάθειες. Μόλις λήξουν οι προθεσμίες, τότε πρέπει κανείς να είναι αργά για το, να ετοιμάσει το δελτίο. Νομίζω ότι για τη διεθνή διάσταση του θέματος έχω ήδη μιλήσει. Ελπίζω λοιπόν ότι απέντησα στις ερωτήσεις, Πρόεδρε, και ότι έχω καλύψει τις ανησυχίες των κλειτών. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ντάνσετ για την παρουσία σας καθώς και για την απάντηση στις, ε, απαντήσεις μάλλον ερωτήσεις. Εκφράστηκαν επιθυμίες σήμερα. Την μεγαλύτερη επιθυμία μας την εκπληρώνεται. Και όπως λένε, αυτός που παραγγέλνει τη μουσική πρέπει και να την πληρώσει κιόλας. Εμείς λοιπόν που σας αναθέτουμε καθήκοντα πρέπει να φροντίσουμε και για τη χρηματοδότησή σας. Βεβαίως να προωθηθούν και άλλα θέματα. Θα είναι ένας διαρκής αγώνας, αλλά βεβαίως η νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος συνεπάγεται και δαπάνες. Εμείς είμαστε η μία πλευρά, η άλλη πλευρά είναι το Συμβούλιο και βεβαίως μαζί τα αποφασίσαμε, τα εγκρίναμε αυτά τα πράγματα ως συνομοθέτες, μαζί πρέπει να εξεύρουμε και την απαραίτητη χρηματοδότηση για τον οργανισμό σας ώστε τα πράγματα τα οποία συζητήσαμε μαζί και τα οποία μας υποσχεθήκατε να μπορέσουν και να υλοποιηθούν. Σας ευχαριστώ. Οφείλω να σας ομολογήσω ότι είμαστε υπερήφανοι για τους οργανισμούς μας. Εξυπηρετούν το σύνολο των 500 εκατομμυρίων κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως Υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία πρέπει να καλύψουν οι οργανισμοί, θα έπρεπε τουλάχιστον. Φαίνεται καθαρά ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο. Ο δρόμος είναι βεβαίως δυσχερής και σπαρμένος με εμπόδια, ωστόσο αξίζει τον κόπο. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ και την εκπρόσωπό μας, του Κοινοβουλίου δηλαδή, που μόλις προσήλθε. Δυστυχώς υπήρξε όπως φαίνεται κάποια παρανόηση για την έλευσή της, αλλά πάντως τώρα είναι παρούσα. Εδώ λίγη η συζήτηση με τον κύριο Ντάνσετ. Εύχομαι καλή επιτυχία στο περαιτέρω έργο σας. So, Ακολουθεί το επόμενο θέμα της ημερησίας διατάξεως που είναι το υπαριθμόν 20 δραστηριότητες του ΣΤΟΑ ή της ΣΤΟΑ σχετικά με την αηφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων. Ο συνάδελφός μας θα κάνει την εισαγωγή, ο κύριος ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Έχοντας αναλάβει την πρωτοβουλία και την εποπτεία του ε, project της ΣΤΟΑΣ για τη διαχείριση των νερών, εκφράζω τις ευχαριστίες μου στην Επιτροπή σας που δέχεται να συζητήσει την προσωρινή έκθεση για τη διαχείριση των νερών. Όταν πρότεινα στο πάνελ της ΣΤΟΑΣ να αρχίσουμε αυτή την ε, ιστορία για την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των νερών. Είχα την αίσθηση και εξακολουθώ να την έχω σήμερα ότι αυτός ο τομέας είναι ο λιγότερο ανεπτυγμένος ε, σχετικά με την αποδοτικότητα των πόρων διότι οι, όσοι ασκούν την πολιτική αλλά και στα μάτια του κοινού η σπατάλη του νερού ίσως ε, παίζει ένα λιγότερο σημαντικό ρόλο από τη σπατάλη της ενέργειας και άλλων πόρων. Στην μελέτη μας αυτή προσπαθούμε να προτείνουμε λύσεις ή να διαγράψουμε κάποιες ενδεχόμενες καλές λύσεις στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη, τουλάχιστον για την ώρα, δεν σημειώνεται κρίση σχετικά με το καθαρό νερό. Υπάρχει όμως σαφώς μια σπάνιδα στις μεσογειακές χώρες. Και στην κεντρική περιοχή της Ουγγαρίας το πρόβλημα που σημειώνεται είναι μεγάλο. 10% του ευρωπαϊκού πληθυσμού θίγεται από την ε, σπάνιδα των νερών. Στην μελέτη αυτή περιλαμβάνω συγκεκριμένη πρόταση ώστε οι συντάκτες της μελέτης όχι μόνο να καταγράψουν την ε, ισχύουσα κατάσταση, αλλά να προτείνουν και λύσεις. Δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε εμείς οι ευρωβουλευτές για, τον τομέα αυτό πρώτα να δούμε ποια είναι τα καλύτερα παραδείγματα, οι πιο καλές πρακτικές στην Ευρώπη. Εδώ έχω δύο παραδείγματα. Αφενός στην Βάδη Βερτεμβέργη, γερμανικό κρατήδιο, όπου ο αγρότης, εάν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν υπάρχουν νητρικά πάνω από 15 μιλιγκράμμ ανά ε, Αναλύτρω λαμβάνει μια ειδική ενίσχυση. Είναι σημαντικό αυτό, διότι ο, η Βάδη Βιρτεμβέργη, το κρατήδιο δηλαδή του Ομοσπονδιακή αυτή η χώρα της Γερμανίας, πληρώνει για τη διατήρηση ενός δημόσιου αγαθού. Άλλο τώρα ε, παράδειγμα, ε, σε ιδιωτική βάση στη Γαλλία. Η ε, γνωστή εταιρεία εμφιαλωμένων νερών Vitel ακολουθεί ένα παρόμοιο σύστημα έχει κάνει μακρόχρονες συμβάσεις με τους αγρότες υπό την ισχύ των οποίων τους προσφέρει 200 ευρώ ανά εκτάριο καθώς και ένα ποσό κατά αποκοπήν αρχικά δηλαδή 150.000 ευρώ για να καλύψουν έτσι το αρχικό κόστος επενδύσεων για τη βελτίωση των τεχνικών διαχείρισης ε, των εδαφών τους. Να λοιπόν, καλές πρακτικές τις οποίες μπορούμε να ακολουθήσουμε. Το δεύτερο θέμα είναι η τεχνολογική ενίσχυση του εξυγχρονισμού. Όχι μόνο, όχι μόνο ε, στην αγροτική οικονομία, αλλά και στη διαχείριση των λιμάτων. Για παράδειγμα, πάρτε το Λονδίνο, όπου ένας εκπρόσωπος Ισραηλινής ε, εταιρείας μου είπε ότι πριν εξυγχρονίσουν ε, τη διαχείριση των ε, αστικών λιμάτων, το 30% κατεσπαλάτο. Δηλαδή ε, χανόταν λόγω τεχνολογικών προβλημάτων. Το άλλο είναι βέβαια και το θέμα της εκ νέου χρήσης, ανακύκλωσης του νερού. Είναι πολύ χαμηλή, χαμηλό το ποσοστό για την ώρα, ενώ σε σύγκριση, σε σύγκριση με το Ισραήλ, όπου 80% των νερών ανακυκλώνονται. Ενώ στην Ευρώπη μόνο η Ισπανία φτάνει το 25% και οι άλλες χώρες είναι πολύ χαμηλότερα. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την, νέα, την εκ νέου χρήση των νερών, εκεί έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε. Τρίτο στοιχείο που αναφέρεται στα κίνητρα. Για παράδειγμα, στην άρδευση. Στα νερά που χρησιμοποιούνται για αρδευτική χρήση δεν υπάρχει ογκομετρική ογκομετρικός υπολογισμός των τιμών. Γιατί, γιατί οι αγρότες δεν έχουν ε, κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ε, μην σπαταλούν το ε, νερό. Νομίζω ότι πρέπει να γίνουν κάποια βήματα και στον τομέα αυτό. Και ποιο είναι το σημαντικότερο συμπέρασμα αυτής της προσωρινής μελέτης. Ότι σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία δεν υπάρχουν κοινέ προδιαγραφές, δεν υπάρχει κοινή ε, νομοθεσία πλαίσιο σχετικά με το πρόβλημα ποιο νερό μπορεί να χρησιμοποιείται για άρδευση και με ποιο επίπεδο επεξεργασίας. Αυτό είναι το μεγάλο εμπόδιο στο ευρωπαϊκό επίπεδο και εγώ νομίζω ότι στον τομέα αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε κάποια πρωτοβουλία στο ευρωπαϊκό επίπεδο διότι η ανακύκλωση του νερού από τη μια μεριά, η εκ νεού χρήση του νερού, αυτά λοιπόν από τη μια μεριά, από την άλλη μεριά να υπάρχουν οι κοινέ προδιαγραφέ στον τομέα αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικές. Επίσης χαίρομαι διότι στο πλαίσιο της κοινή αγροτική πολιτικής, της μεταρρύθμισης τη ΚΑΠ δηλαδή, το λεγόμενο greening, το πρασίνισμα δηλαδή, παίζει πλέον ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Στον δεύτερο πυλώνα θα εγγραφούν κονδύλια για τον εξυγχρονισμό των αρδευτικών συστημάτων στην Ευρώπη. Αυτό το βρίσκω πολύ σημαντικό. Έχω καταθέσει και μια σχετική τροπολογία, διότι γινόταν βέβαια κάποια διάκριση υπέρ των παλαιών χωρών μελών. Εγώ είπα λοιπόν με την τροπολογία μου και οι παλαιές και οι νέες χώρες μελή να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα αυτά, τα κονδύλια αυτά για τον εξυγχρονισμό των αρδευτικών συστημάτων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Η Σάντρα Μπέρμαν. Θα σας παρουσιάσω τα αποτελέσματα τα ενδιάμεσα αποτελέσματα από την ε, μελέτη του πάνελ ΣΤΟΑ για την ε, βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων με ειδική εστίαση στο νερό και στη γεωργία. Το IEP, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής Πολιτικής, ε, που εκπροσωπείται από την κυρία Πανάκοβα σήμερα, συμμετείχε και το Ecologic. Ε, διτή είναι η εστίασή μας, ε, καταρχάς να εστιάσουμε στην διαχείριση του νερού ως φυσικό πόρο. Όπως είπε ο κ. Σταμπάτζη, ε, το νερό είναι ένα πολύ πολύτιμο φυσικό είδος, φυσικό, ε, φυσικός πόρος για τον άνθρωπο και η διαχείριση των φυσικών πόρων που συνδέονται με την ε, Ευρωπαϊκή Γεωργία. Φυσικά υπάρχουν πολλές σχέσεις μεταξύ των δύο στόχων, γιατί το νερό είναι μια πολύ σημαντική πηγή για την γεωργία και η γεωργία έχει πολύ σημαντική επίπτωση στο νερό και θετική και αρνητική. Στο πρώτο τμήμα της διαχείρισης του νερού ε, εξετάζουμε το ρόλο της έρευνας, της τεχνολογίας, των βέλτιστων πρακτικών για την αποτελεσματική και αποδοτική χρήση του νερού. Ε, τα ωφέλη, τα αντισταθμίσματα, για το έδαφος, για το νερό, για τον αέρα, συγγνώμη, και για τα κατάλοιπα και να δούμε ε, τι υποστήριξη χρειαζόμαστε μέσω της ΚΑΠ ή μέσω άλλων χρηματοδοτικών μέσων. Στον αγροτικό τομέα, στο αγροτικό σχέλος, ε, βλέπουμε τι επιλογές έχουμε για την διαχείριση του εδάφους, ε, τη σχέση με την κλιματική αλλαγή και τι επιλογές έχουμε για να διασφαλίσουμε την, να μην προωθήσουμε την κλιματική αλλαγή. Επίσης, μέτρηση του νερού και έχουμε εστίαση στα αγροπεριβαλλοντικά θέματα. Για τη χρήση του νερού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να σας δείξω το πλαίσιο της προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη σε σχέση με το νερό, έχετε αυτό το μικρό διάγραμμα που δείχνει ότι το περισσότερο νερό χρησιμοποιείται για την παραγωγή ενέργειας, το νερό που αντλούμε, έτσι. Γιατί άλλο η άντληση και άλλο η κατανάλωση και το 22% του νερού χρησιμοποιείται από τη γεωργία κατά μέσο όρο. Όμως είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι η μεγάλη διαφορά στα κράτη-μέλη, πάνω από το 80% το νερού χρησιμοποιείται στην Ισπανία για την άρδευση Ενώ η έλλειψη αφορά κυρίως τα νότια κρατή μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά παρόλα αυτά, ε, στην ε, κεντρική Ευρώπη, γύρω από τα ποτάμια, αλλά και στο νότιο-ανατολικό Ηνωμένο Βασίλειο, και είναι ένα θέμα που πρέπει να ληφθεί υπόψη γενικά πολύ σοβαρά και στα άλλα κράτη-μέλη γιατί υπάρχει σχέση ανάμεσα στο νερό και στην ενέργεια. Όταν χρησιμοποιείς νερό, ε, χρησιμοποιείς ενέργεια για την άντληση, για την επεξεργασία, για τη θέρμαση κτλ. Και η κλιματική αλλαγή αναμένεται να ε, επιδεινώσει τα σχετικά προβλήματα. Οι τέσσερις προκλήσεις στην Ευρωπαϊκή Γεωργία είναι η ύπαρξη, η διαθεσιμότητα νερού. Στον αγροτικό τομέα, ας πούμε, χρησιμοποιείται για την άρδευση το νερό, αλλά αλλά για την κτηνοτροφία και για την μεταποιητική αγροτική βιομηχανία. Η ποιότητα του νερού είναι η δεύτερη πρόκληση, ε, η μόλυνση που υπάρχει γενικά, διάχυτη, ε, οι ροές των υδάτων ε, στους ποταμούς μέσω το, της άρδευσης και τέλος η γεωργία έχει και μία συνιστόσα που αφορά το έδαφος επηρεάζει τις υδάτινες ροές, ε, εξαρτάται, επηρεάζει τη δίθηση, τα ποσοστά δίθησης και μέσω της συζηματοποίησης ε, μολύνει και το νερό. Η κατάσταση του εδάφους δηλαδή. Περισσότερες ε, λεπτομέρειες τώρα για τη διαχείριση του νερού. Πρώτο τμήμα. Εξετάζουμε στην επιστημονική έρευνα που έχουμε και τι βρήκαμε, ότι οι περισσότερε πρωτοβουλίε που αφορούν την αποτελεσματική αποδοτική χρήση του νερού στην Ευρώπη μιλούν κυρίω για τι τεχνικέ άρδευση, καταρχά στην μεταπητική βιομηχανία και στη γεωργία και πώ μπορούμε να συλλέξουμε στοιχεία για να καταλάβουμε καλύτερα τι ανάγκε στη γεωργία. Υπάρχει μια εστίαση στην ολοκληρωμένη διαχείριση των δάτινων πόρων και στην ενισχυμένη συνεργασία, οριζόντια και κάθετα, δηλαδή μεταξύ των διαφόρων χρηστών του υδάτου, αλλά και σε διάφορα, διάφορες κλίμακες, α, ποτάμιες, λεκάνες κτλ. Έρευνα γίνεται σε επίπεδο οικονομικών μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας και διαχείριση στην, στις αστικές περιοχές και στη βιομηχανία. Υπάρχουν κενά σε ό,τι αφορά την ποσότητα του νερού, ε, τις οικολογικές ροές, δηλαδή ροές που πρέπει να παραμείνουν στους ο, όγκους, στους δεξαμενές, ούτως ώστε να υπάρχει διατήρηση της βιοπικιλότητας κτλ. Υπάρχουν πολλές προσπάθειες που μπορούμε να κάνουμε για να υποστηρίξουμε την αποδοτική χρήση του νερού. Οι προτεραιότητες, οι ερευνητικές είναι να δούμε τι, διά, υπόλοιπα νερού έχουμε, ποια είναι η λειτουργία του εδάφους ε, και ποια είναι η ποιότητα του νερού. Οι τεχνολογίες που έχουμε στη διάθεσή μας. Το πρώτο πόρισμα είναι ότι έχουμε πολλές δυνατότητες ε, για αποτελεσματική χρήση του νερού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όλες ε, είναι επωφελείς και προσαρμοσμένες για τις διάφορες περιοχές και τα διαφορετικά αγροτικά συστήματα που έχουμε στην Ευρώπη. Προσπαθούμε να κατηγοριοποιήσουμε αυτές τις επιλογές. Έχουμε 7 διαφορετικές κατηγορίες. Ε, παρακολούθηση της χρήσης του νερού με τη μέτρηση. Ε, μέτρα αξιολόγησης, ε, παραδείγματο χάρη διάφορα αποτυπώματα. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Εταιρική Σχέση που δίνει πιστοποίηση, τεχνολογίες μεταφοράς, καναλιζάρισμα για να μειώσουμε την απώλεια του νερού, Υπάρχουν ε, συγκεκριμένες ε, τεχνικές άρδευσης, τριπλή άρτευση, εναλλακτικές χρήσεις μέσω δεξαμενών κτλ, ε, δυνατότητες διαχείριση μέσω της γεωργίας, κατάλληλες καλλιέργειες, κατάλληλες περιοχές και θέματα χρηματοδότησης. Διερευνήσαμε επίσης τεχνολογίες με την αποτελεσματική μεταφορά με σένσορες κτλ. Καλές πρακτικές. Κοιτάξαμε τις περιοχές υπαίθρου αλλά και τις αστικές περιοχές και τη σχέση ανάμεσα στις δύο. Ε, Παναχρησιμοποίηση των λιμάτων είναι πολύ σημαντικό και είναι σημαντικό οι πολιτικές να εφαρμόζουν κάποιες δράσεις και όλες οι τεχνολογίες αυτές που είπαμε να εφαρμόζονται μέσω κατάλληλων πολιτικών. Η τιμολόγηση επίσης θα πρέπει να απεικονίζεται μέσω διαφορετικών πολιτικών. Ε, σημαντική είναι να υπάρχει και μια στρατηγική προσέγγιση ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε ότι λαμβάνουμε τα πάντα υπόψη, τα σύνα εκτιμούμε όταν αποφασίζουμε για μια συγκεκριμένη πολιτική. Κυρία Πέρμαν, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση του θέματος και θα παρακαλέσω ευθύς αμέσως την κυρία Πολάκοβα να λάβει το λόγο που είναι εκπρόσωπος του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Πολιτικής για θέματα περιβάλλοντος. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα συνεχίσω την παρουσίαση Στο σημείο τομής, δηλαδή θεμάτων διαχειρίσεως νερού και της αγροτικής οικονομίας, εκεί δηλαδή όπου είναι το interface των δύο, ε, των δύο ερευνών, είναι και θέματα διαχειρίσεως ε, γεών, που είναι σημαντικό για το νερό. Αν εφαρμοστούν σωστά, η διαχείριση του εδάφους δηλαδή, μπορεί να αποφέρει σημαντικά ωφέλη. Διατηρεί και βελτιώνει τη λειτουργικότητα του εδάφους καθώς και την ικανότητα του εδάφους ε, να προσφέρει και υπηρεσίες στα οικοσυστήματα, για παράδειγμα με τη συγκράτηση των νερών μακροπρόθεσμα. Αυτά μπορούν να βοηθήσουν και την καλύτερη ανθεκτικότητα των οικοσυστημάτων και επομένως να συγκρατήσουν και τις κλιματικές αλλαγές. Ταυτόχρονα το έδαφος μπορεί να συγκρατήσει και το διοξείδιο του άνθρακα. Αυτό γίνεται σιγά σιγά γνωστό. Λιγότερο συχνά, ωστόσο, τονίζεται ότι τις τελευταίες δεκαετίες μεγάλα τμήματα των ευρωπαϊκών εδαφών έχουν γίνει πηγές ε, ρήπων λόγω της χρήσης ε, των ε, ε, ε διοκτώνων, ζητανιοκτώνων κλπ. αλλά και λόγω των κλιματικών ε, επιρών, Άρα υπάρχει σημαντικό δυναμικό εφόσον γίνει σωστή διαχείριση να μειωθούν αφενός αυτές οι εκπομπές, ταυτόχρονα να διατηρηθεί η ε, δυνατότητα συγκράτησης διοξιδιού άνθρακα όπου αυτή υπάρχει. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Οι επιλογές για την διαχείριση του εδάφους έχουν ορισμένες επιλογές. Είναι σημαντικό να αντιληφθεί κανείς ότι είναι σημαντικό για τη διαχείριση του είναι σημαντική η διαχείριση του εδάφου, για να επιτευχθούν ορισμένοι στόχοι ε, περιβαλλοντικοί, για παράδειγμα διατήρηση ε, αποθεμάτων νερού. Χρησιμοποιώντα για παράδειγμα φυτικά είδη τα οποία αντέχουν στην ξηρασία να, διατηρηθεί η, ε, να διατηρηθούν υπόγεια ύδατα μείωση της ανάγκης σε, νερά διαφόρων καλλιεργιών. Υπάρχουν και άλλοι στόχοι, υπάρχουν και άλλοι τρόποι μάλλον για να υλοποιηθούν οι στόχοι. Ίσως και υπάρχουν και κάποιες συνέργειες με την διαθεσιμότητα νερών, αλλά δεν υπάρχουν πάντα τέτοιες συνέργειες. Εάν στοχεύσουμε την διαχείριση των εδαφών για την επίτευξη στόχων, αυτή θα προσφέρει και σημαντικά ωφέλη και στην προσαρμογή. Εμείς εξετάσαμε όλες τις επιλογές αυτών των ε, στόχων διαχείρισης. Έχουμε περίπου 15. Θα τα βρείτε αυτά βεβαίως και στην προσωρινή μας έκθεση. Ξεκινούμε από απλά μέτρα. Βάζουμε δηλαδή κάποια, κάποιες ζώνες ε, ανακοπής των ε, buffers buffer strips δηλαδή ναι, ορισμένες τεχνικές οργώματος, τρόπους ε, διατήρησης ή αποκατάστασης ε, υγροτόπων, ε, επίσης άλλα μέτρα με τα οποία θα βελτιώσουμε στις επόμενες φάσεις. Και έρχομαι στην επόμενη φάση της μελέτης αυτής που είναι η κοινή αγροτική πολιτική. Κάναμε δουλειά για να εντοπίσουμε τις διάφορες τάσεις οι οποίες επηρεάζονται από τη γεωργία και που επηρεάζουν τη γεωργία. Δεν θα τα πω όλα αυτά εδώ. Ίσως ε, γνωρίζετε ότι υπάρχουν θέματα, αυτά δηλαδή που ανέφερε ο κ. Νταμπάζδη ήδη για την ε, ύπαρξη για τη διαχείριση των νερών θέματα, για τη ε, διαχείριση των ροών ποταμών και συνέργειες με τη διαχείριση του εδάφους. Θα βρείτε πολλές λεπτομέρειες στην προσωρινή έκθεση. Τώρα, να σας εξηγήσω την ανάλυση μας για τα μέτρα υπό την ισχύ της κοινή αγροτικής πολιτικής. Εδώ υπάρχει ένα φάσμα μέτρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το νερό και στον πρώτο και στο δεύτερο πυλώνα. Μεταξύ αυτών η πολλαπλή συμμόρφωση και το μέτρο αγροτικού περιβάλλοντος, agri environment, που είναι σημαντικά για τα νερά στην Ευρώπη. Υπάρχουν όμως και άλλα μέτρα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορους ε, σκοπούς και θα σας τα εξηγήσω. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι δεν υπάρχει σαφήνεια σχετικά με τα ποια ε, κοινοτικά ταμεία ε, πηγαίνουν για την διατήρηση των νερών λόγω των διαρθρώσεων. Είναι δύσκολο λοιπόν να βρεθούν τα σωστά στοιχεία για τα ταμεία τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για χρηματοδότηση έργων για τα νερά. Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν και θέματα αποτελεσματικότητας όλων αυτών των μέτρων στον πρώτο και στον δεύτερο πυλώνα. Θα ήθελα να, ρίξουμε ιδιαίτερη, να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στα αγροτοπεριβαλλοντικά μέτρα, τα οποία είναι κρίσιμα διότι επιτρέπουν την στόχευση και την διαμόρφωση των ε, μέτρων έτσι ώστε να εξυπηρετούν τους στόχους αυτούς σε διάφορα περιβαλλοντικά θέματα, για παράδειγμα ειδικότερα για το νερό, αλλά και το νερό, οι ανάγκες του νερού μπορεί να είναι διαφορετικές από μια χώρα ε, σε άλλη αλλά και από μια περιφέρεια σε άλλη. Είναι λοιπόν σημαντικό να ε, φτιαχτούν μέτρα τα οποία να στοχεύουν σε ειδικέ ε, ανάγκες. Για την περίοδο 2007 έως 2013 που είναι αυτή που μας απασχολεί, οι management actions έχουν διαφορετικούς στόχους σε ό,τι αφορά την ποιότητα των νερών, τις ροές, την διαθεσιμότητα νερού και τις λεγόμενες cross-cutting actions, που περιλαμβάνουν και θέματα διοίκησης, διαχείρισης, τα οποία θα σας εξηγήσω σε λίγο. Το κέριο ερώτημα είναι όχι μόνο πώς χρησιμοποιήθηκαν τα μέτρα αυτά από τις χώρες μέλη, αλλά και πώς, πώς αποτελεσματικά είναι για την προστασία των νερών. Εμείς έχουμε ε, συλλέξει πολύ άριθμα παραδείγματα συγκεκριμένων ε, προγραμμάτων σε πολλές χώρες μέλη τα έχουμε ταξινομήσει ανά θέματα. Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν την ωφέλεια τέτοιων προγραμμάτων, ιδίως για την μείωση της χρήσης ε, ζυζανιοκτώνων και λιπασμάτων. Υπάρχει ένα θέμα στα, στα ρώσιμες Υπάρχει ένα θέμα με τις γενικευμένες ε, πληρωμές για την μείωση των λιπασμάτων, γιατί υπάρχει μια δυσκολία να μετρηθούν οι άμεσες επιπτώσεις στο νερό αυτών των ε, πληρωμών. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχει θέσει και το ελεγκτικό συνέδριο πέρσι στην έκθεσή του. Άλλο θέμα είναι ότι οι ενδείξεις που έχουμε για τις πραγματικές επιπτώσεις στα νερά είναι πολύ περιορισμένες λόγω της περιπλοκότητας των στόχων, λόγω των περιορισμένων δεδομένων και επίσης διότι οι τάσεις για τη βελτίωση των νερών είναι μακροπρόθεσμης εξέλιξης μέχρι δηλαδή να γίνουν ορατές. Δεν υπάρχουν τόσο πολλές μελέτες οι οποίες να μπορούν να μας βοηθήσουν να αξιολογήσουμε την πραγματική βελτίωση των νερών. Ορισμένα θέματα, όπως και η αποτελεσματικότητα των αγροτοπεριβαλλοντικών μέτρων, προκύπτουν και από ασθενείς στόχους, όπως εξήγησα και προηγουμένως. Ένα παράδειγμα είναι όταν δίνουμε γενικευμένες πληρωμές για να μειώσουμε τις επιπτώσεις, για παράδειγμα, στη διάβρωση των εδαφών, αλλά δεν είναι στοχευμένες ειδικά στις περιοχές όπου προκύπτουν τα προβλήματα αυτά. Αυτό είναι κάτι άλλο το οποίο συνεπέρανε, το οποίο σημείωσε το ελεγκτικό συνέδριο στην έκθεσή του, αλλά έχει και άλλα παραδείγματα πέρα από τα αγροτοπεριβαλλοντικά μέτρα τα οποία μπορεί να καλύπτουν πληρωμές για διάφορα είδη διαχείρισης των εδαφών υπάρχουν και κεφαλαιοχικές επενδύσεις στον πυλώνα 2 στην, ε, στις υποδομές δηλαδή για την βελτίωση των νερών. Τα μέτρα αυτά για το 2007 έως 2013 είναι υποδομές για την προσαρμογή της γεωργίας, μη παραγωγικές επενδύσεις και ούτω Όλα αυτά τα μέτρα διατηρούνται στην πρόταση για τη μελλοντική κοινή αγροτική πολιτική με κάπως διαφορετικούς τίτλους, αλλά στην βάση τα μέτρα αυτά, όπως είπα, διατηρούνται. Οι σκοπούμενες βελτιώσεις αυτών των επιχορηγήσεων είναι, για παράδειγμα, για να βελτιωθεί η διαδεσιμότητα των νερών, που υποτίθεται ότι θα επιτευθεί με την λήψη δράσεων που στοχεύουν στην εκ νέου χρήση των νερών, για παράδειγμα τη συλλογή των βρόχινων νερών στις ε, εκμεταλλεύσεις και ε, μείωση της ανάγκης άρδευσης. Υπάρχουν και ε, άλλες επιπτώσεις, για παράδειγμα με, την, με επενδύσεις στον εξυγχρονισμό των αποχετευτικών συστημάτων. Υπάρχουν όμως και ορισμένα ερωτήματα που τίθεται από την περιβαλλοντική σκοπιά σε σχέση με αυτές τις επενδύσεις πολύ λίγα στοιχεία διαθέτουμε σχετικά με τις επενδύσεις που γίνονται για την άρδευση, εάν δηλαδή όντως έχουν οδηγήσει σε εξοικονόμηση νερών. Δεν γνωρίζουμε. Για τα αποχετευτικά συστήματα, πολλοί που ε, γνωρίζουν ποια είναι τα αποτελέσματα των, των, των αποχετευτικών συστημάτων, κατανοούν ότι υπάρχουν και μεγάλοι κίνδυνοι που συνδέονται με την ε, Έτσι λοιπόν είναι απαραίτητο να συλλεχθούν στοιχεία, διότι αυτή τη στιγμή λείπουν. Στο επόμενο βήμα εμείς θα ε, κάνουμε πιο λεπτομερή αξιολόγηση, θα ε, προτείνουμε και policy options και θα ε, συνδέσουμε τις, ε, μελέτη, τη μελέτη μας και με το σχέδιο της Κομισιόν το οποίο πρόσφατα δημοσιεύτηκε. Και αυτά για τον επόμενο Μάρτιο μέχρι Μάιο. Ευχαριστώ. Τα Ταρέλα και μετά Πρόντι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που προβλέψατε στην ημερήσια διάταξη αυτά τα δύο θέματα και τις παρουσιάσεις. Μου δίνετε την ευκαιρία να θέσω μια ερώτηση μεθοδολογίας. Αυτή τη στιγμή είχαμε ένα πολύ μικρό απόσπασμα από το εξαιρετικό έργο που κάνει στο Το πρόβλημα είναι το εξής. Πώς να γίνει ακόμα χρησιμότερη και εξυπηρετική η όλη δράση της ΣΤΟΑ. Πολλές φορές έχω την εντύπωση ότι όσα κάνει η στόα γίνεται κάπως σαν αυτοσκοπός εκτός από κάποιες εξαιρέσεις όπως η σημερινή αλλά δεν φαίνεται να αξιοποιούνται οι έρευνες της ΣΤΟΑ στην Επιτροπή μας, κατά κύριο λόγο, και σε άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Θα πρέπει λοιπόν να ζητήσουμε έναν τρόπο, διότι είναι κάτι που καθημερινώς το αντιμετωπίζουμε. Έχουμε τεχνικά προβλήματα και επιστημονικά προβλήματα πολύ συγκεκριμένα καθημερινά. Γιατί και αυτό πολλές φορές μας αναγκάζει να παραδεχτούμε την μη πλήρη γνώση ενός αντικειμένου. Συχνά επίσης είμαστε θύματα ε, ομάδων ασκή, άσκησης πίεσης που μας τραβάνε από το γιακά και προσπαθούν να μας πείσουν για διάφορα πράγματα. Ή στο άλλο λοιπόν, εφόσον έχει ανεξάρτητους ερευνητές που εκπονούν ε, μελέτες, θα μπορούσε ως όργανο και ως μέσο να μας χρησιμεύσει σαν ένα πιο αξιόπιστο και λιγότερο μεροληπτικό εργαλείο γνώσης από ότι ομάδες άσκησης ε, πίεσης. Εδώ ούτε την ε, στο εκπροσωπώ, ούτε ανήκω σε κάποια ομάδα για την οποία, μέρος της οποίας ε, μιλώ, ούτε τον εαυτό μου. Την κοινοβουλευτική μας επιτροπή εκπροσωπώ. Εδώ λοιπόν, εφόσον το Προεδρείο έχει αναθέσει συγκεκριμένες αρμοδιότητες ε, στις διάφορες επιτροπές και εφόσον εμείς έχουμε τόσο σοβαρά ζητήματα να εξετάσουμε, μπορούμε να απευθυνόμαστε στη ΣΤΟΑ και να ζητούμε την εκπόνηση μελετών, ε, αναλύσεων, ε, οργάνωση εργαστηρίων και σεμιναρίων. Από κοινού τη ΣΤΟΑ έχουμε οργανώσει και κάποια workshop με ε, συμμετοχή εξαιρετικών επιστημόνων. Δυστυχώς όμως, σε αυτές τις περιπτώσεις, η, η έλευση των ε, συναδέλφων βουλευτών που έχουν προσκληθεί παρόλα αυτά και επανειλημμένως, δεν είναι σταθερή, ούτε αρκετή. Θα πρέπει απλώς να αξιοποιήσουμε καλύτερα το έργο της ΣΤΟΑ στο μέλλον. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κύριε κύριος Πρόντι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για την ευκαιρία. Θα συμφωνήσω με ως υποσυνάδελφος Ταταρέλα και θα δώσω και μια συνέχεια, γιατί εγώ εκπροσωπώ την Επιτροπή Ένβη στη ΣΤΟΑ ακριβώς. Άρα Είμαι ο ίδιος επιφορτισμένος με την εξέταση κάποιων θεμάτων. Προσπαθούμε να καλύψουμε κάποια κενά τα οποία προέκυψαν και στην όλη μας συζήτηση. Πιο συγκεκριμένα. Αυτή τη στιγμή τη συζητάμε. Τεχνολογικά μέσα και λύσεις για το πώς θα εξασφαλίσουμε την ε, τροφή για δέκα ε, ανθρώπους. Την νανοασφάλεια, θέματα τοξικολογικά που σχετίζονται με μόρια τα οποία ορούνται στο νερό και πρέπει να μπορούν να μετρηθούν από τα λεγόμενα νανόμετρα. η διάμετρός τους δηλαδή. Υπάρχουν επίσης επιστημονικά ζητήματα, με μεθεντολογικές διαστάσεις και ηθικές θα πρέπει να σκεφτούμε ας πούμε το ανθρώπινο DNA, το γονιδίωμα ή το making perfect life και human ε, enhancement, ε, για την κλωνοποίηση ακόμη. Αυτά δείχνουν πόσο σημαντικό εργαλείο μπορεί να είναι η για το Κοινοβούλιο. Θα έχετε ακούσει όλοι ότι ο πρόεδρος Μπαρόζο έχει έχει αναθέσει επιστημονικές αρμοδιότητες και υπάρχει επιστημονικός επιτετραμένος ε, παρά το κ. Μπαρόζο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, αυτά απλώς να πω ότι είμαι στη διάθεσή σας για περαιτέρω συζητήσεις, γιατί και η σημερινή ανταλλαγή απόψεων είναι χρήσιμη και γι' αυτό θέλω να παρέμβω στο θέμα της συγκεκριμένη μελέτης, ιδίως για τα είδατα. Πρέπει να έχουμε ως προτεραιότητα κατά νου το πρόβλημα της προσαρμογής μας στις κλιματικές αλλαγές. Το νερό. Το νερό είναι κομβική σημασία για το σκοπό αυτό. Εάν θέλουμε να διαφυλάξουμε τα εδάφη μας, πρέπει να σκεφτούμε τι θα γίνει με την κατακράτηση υδάτων. Οι βροχοπτώσεις είναι πιο έντονες αλλά λιγότερο συχνές. Θα πρέπει λοιπόν να κατακρατείτε το νερό εκεί που έχει πέσει μέσα από την βροχή όσο το δυνατόν περισσότερο. Υπάρχουν και, τα λεγόμε, και οι υδροφόροι ορίζοντες εδώ που θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ο σύστημα διαχείρισης των υδάτων. Επίσης θα μπορούσαμε να δούμε πώς θα αντιμετωπίζουμε τις πλημμύρες ε, σε όλο αυτό το πλαίσιο. Το νερό είναι ένα ολόκληρο πολύπλοκο σύστημα. Υπάρχουν παράμετροι που σχετίζονται με το νερό που μπορεί να έχουν και πολύ θετική, χρήση. Ο φόσφορος λόγου χάρη. σε περίπου 50 χρόνια θα υπάρχει έλλειψη του στοιχείου αυτού. Κάποιες φορές υπάρχει και υπερβολική χρήση του στοιχείου στην ε, Γεωργία. Το πρόβλημα λοιπόν είναι το εξή. Πώ θα διαχειριστούμε το νερό κατά τρόπο τέτοιο, ώστε ιδίω για τα αστικά κέντρα, τι αστικέ περιοχέ, να ανακτήσουμε το οργανικό αυτό κομμάτι που από την άλλη θα μπορούσε να αξιοποιείται για ιατρικούς σκοπούς, για ενεργειακούς σκοπούς μάλλον, και τα σύνθετα μέρη του να αξιοποιούνται στη γεωργία. Αυτά όλα λοιπόν πρέπει να διαφυλαχθούν. Ιδιαιτέρως για τα αστικά κέντρα, η επεξεργασία των υδάτων και των λιμάτων περιλαμβάνει διαφορετικές πτυχές. Έχουμε διαφορετικές περιπτώσεις. Να θυμίσω το εξή. Τα ύδατα από τις, τα λίματα από τις αποχετεύσεις θα μπορούσαν να τύχουν επεξεργασίας και να αξιοποιηθούν και έτσι να επιστρέφει το νερό καθαρισμένο πλέον στους υδροφόρους ορίζοντες. Και εδώ πραγματικά υπάρχουν ε, συμπτώσεις και συγκυρίες φαινομένων φυσικών που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και να αποβούν προς όφελός μας. Θα πρέπει λοιπόν την μελέτη αυτή να την δούμε συνολικά, για να, σφαιρικά μάλλον και με απόσταση, για να αντιληφθούμε το νερό σύστημα ως σύστημα με πολλές συνιστώσεις. Κάτι που έγινε στο Αμβούργο λόγω χάρη, σε μια συνοικία του Αμβούργου στη Γερμανία. Με ακάθαρτα ύδατα με μεγάλη ποσότητα οργανικών ουσιών οι οποίες θα μπορούσαν να αποσπαστούν και μετά να αξιοποιηθούν στην παραγωγή ενέργειας. Και τα ιχνοστοιχεία, τα ε, οργανικά στοιχεία που θα παραμείνουν να μπορούν και πάλι να χρησιμοποιηθούν. Βλέπετε ότι δημιουργείται ένας κύκλος έτσι. Από τη μια έχουμε την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, την διαφύλαξη των εδαφών και την προστασία τους και από την άλλη το πρόβλημα ανάκτησης υλικού και υλικών με την αντιμετώπιση ενδεχόμενων ελλείψεων. Να λοιπόν, αυτό θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε ως προειδοποίηση και ως μια ευκαιρία για να αντιληφθούμε ότι τίποτα δεν πρέπει να πάει χαμένο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόντι. Ευχαριστώ επίσης πρώτα για την ε, παρουσίασε τις δύο ειδήμονες, η κ. Ταταρέλα και Πρόντι αναρωτήθηκαν πώς μπορούμε να εντάξουμε καλύτερα το έργο της ε, ΣΤΟΑΣ στο έργο της ε, Επιτροπής Περιβάλλοντος, πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή καλύτερα τις εκθέσεις σας για, στην, τεχνική μας, στην καθημερινή μας τεχνική εργασία. Θα παρακαλέσω τους εκπροσώπους των δύο μεγάλων πολιτικών ομάδων να γίνουν προτάσεις πρωτίστως από τις πολιτικές ομάδες. Την ε, συνάντηση των συντονιστών. Να μπορέσουμε τότε να τη συζητήσουμε ενδεχομένως αποδοχή των προτάσεων αυτών ή ενδεχομένως τροποίησή τους, πώς μπορούμε δηλαδή να φροντίσουμε ώστε οι εργασίες της ε, ΣΤΟΑΣ να εμπλουτίσουν την δική μας εργασία, διότι εσείς κάνετε πραγματικά πολύ και καλή δουλειά και είναι σωστό να ε, προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο. Ε, έχω ήδη... Είναι γι' αυτό το θέμα της μεσαίας διατάξεως το επόμενο. Τότε θα πρέπει να ε, δώσω το λόγο και ως σε όλους τους υπολείπους. Δεν προλαβαίνουμε αλλιώς με την προφορική ερώτηση. Προτείνω να μιλήσεις με την Εύελιν που είναι η συντονίστρια ώστε οι προτάσεις να γίνουν στο πλαίσιο των συντονιστών. Ευχαριστώ και πάλι για την συζήτηση καθώς και για την παρουσίασή σας και προχωρώ στο επόμενο θέμα της ημερησίας διατάξεως όπου τον λόγο λαμβάνει αποκλειστικά η κυρία Λίντα Μακάβαν αφού πρόκειται για την προφορική ερώτησή της 2012-08 για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και κυρίως για τα οξύδια του αζότου. Έχουμε εδώ πέρα τους ειδικού της ΣΤΟΑ και θα μπορούσαν να έρθουν σε επαφή με τους εισηγητές να αναλάβουν δράση. Εμείς κάνουμε καλές ε, εκθέσεις, απλώς τις δημοσιεύουμε όμως. Καλό είναι τις, ε, να έρθει σε επαφή, με τους εισηγητές, να δείτε τις εκθέσεις, γιατί φοβάμαι ότι αυτή η καλή δουλειά θα πάει χαμένη. Δεν θα τη δει κανένας καλό είναι να κινητοποιούμαστε και οι μεν και οι δε. Και εμείς στο Κοινοβούλιο και εσείς. Μη φοβάστε λοιπόν να έρθετε σε επαφή ε, απευθείας με τους ε, ευρωβουλευτές. Γιατί αλλιώς γίνεται όλη αυτή η έρευνα ε, και μετά δεν αναφερόμαστε καθόλου σε αυτήν. τώρα, συνήθως για τέτοιου είδους ερωτήσεις δεν ξέρω αν δίνουμε το λόγο στην Κομισιόν. Μιλάμε για την ποιότητα του αέρα. Η Κομισιόν έκανε μια ανάλυση για το πώς τα κράτη-μέλη ε, υλοποιούν τους ε, στόχους ποιότητας. Κάποια κράτη-μέλη και πόλεις μέσα σε κράτη-μέλη προσπαθούν να σεβαστούν αυτούς τους ε, στόχους ποιότητας του αέρα. Το ερώτημα των πολιτών είναι γιατί. Γιατί, γιατί τα κράτη-μέλη και οι πόλεις δεν εφαρμόζουν τα νομοθετήματα, δεν είναι αρκετά αυστηροί στόχοι γιατί κάποιες ε, κυβερνήσεις και κάποιες τοπικές αρχές, όπως λένε, το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει πρόοδος ε, στα οχήματα και στα τεχνικά πρότυπά τους και αυτό δημιουργεί το πρόβλημα. Και κάποια δημοτικά συμβούλια δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Αν ας πούμε τα όρια των εκπομπών είναι πολύ ψηλά. Ε, έχουμε πολιτικές για να ενθαρρύνουν ανθρώπους να αγοράσουν αυτοκίνητα diesel. Εν πάση περιπτώσει, η Κομισιόν πού, έχει φτάσει με την ανάλυση της για τη συμμόρφωση με την οδηγία και ποια κατά την άποψή της είναι τα μείζωνα προβλήματα. Υπάρχει τον επόμενο Ιούνιο ε, μία αναθεώρηση για την ποιότητα του αέρα. Θα γίνει. Και πότε η ανάλυση σας για τη συμμόρφωση των κρατών μελών θα ενσωματωθεί στη νέα νομοθεσία. Ε, θα προτείνετε επίσης νέα πρότυπα ή όχι. Ευχαριστώ. Την Λίντα Μακάβαν. Ε, η Κομισιόν παρακαλώ. Thank you. Good morning, Ευχαριστώ και καλημέρα κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί βουλευτές. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Τόμας Είμαι τμήματάρχης και ασχολούμαι με την ε, ποιότητα του αέρα, με βιομηχανικές εκπομπές και με θόρυβο. Είδα την ερώτησή σας, εσείς τη συνοψίσατε λιγάκι διαφορετικά από ό,τι μας την είχατε υποβάλει. Θα προσπαθήσω αυτό που είπατε όμως να το απαντήσω. Θέλω να σε επιβεβαιώσω ότι η Κομισιόν έλαβε τα δεδομένα για το 2011 για την ποιότητα του αέρα από όλα τα κράτη-μέλη πλέον και όντως υπάρχουν πολλά κράτη-μέλη που παραβιάζουν τις οριακές, τιμέ, τις ε, οριακές τιμές για τα αιωρούμενα σωματίδια. Οι καθημερινές τιμές είναι για τα αιωρούμενα σωματίδια και για τα οξύδια του αζότου είναι ετήσιες οι τιμές. Ε, έχουμε ζώνες ποιότητας αέρα. Όχι με, δεν δουλεύουμε με εθνικά, εθνικές επικράτειες. Είχαμε 250 από τις 650 που ξεπερνούσαν την οριακή τιμή των 10 ppm. Ε, και ένα διαφορετικό νούμερο για την υπέρβαση των ε, οριακών τιμών για το οξύδιο του αζότου. Για το διοξείδιο του αζότου θέλουν επέκταση της προθεσμίας και σήμερα έχουμε λάβει γνωστοποίησεις από 18 κρατημέλη που καλύπτουν 202 ζώνες. Τα διοξίδια του αζότου ε, κλείονται λόγω εξατμίσεων αυτοκινήτων, σχεδιάζονται δηλαδή με την κυκλοφορία, όχι μόνο με την κυκλοφορία, αλλά και με, τις, ε, με τους, βενζιλο, βεν, διζελοκινητήρες. Συγγνώμη. Κάποια κρατημέλη είπαν ότι για 8 ζώνες δεν θα μπορέσουν να σεβαστούν ε, τις τιμές μέχρι το 2020 Ε, θέλουμε να αποφασίσουμε καταρχά για την επέκταση όμω προθεσμία και επομένω ε, δεν το λαμβάνουμε αυτό υπόψη. Έχουμε 9 μήνε για να λάβουμε απόφαση για τι ε, επεκτάσει προθεσμία. Έχουμε μέχρι στιγμή αποφασίσει για τι μισέ ζώνε που εντοπίστηκαν. Ε, κάποιες παραβιάσεις. Για τις 45% δεν έχουμε εκφράσει αντιρρήσεις, γιατί συμμορφούνται τα τα κρατημέλη με τα κριτήρια της οδηγίας και έχουμε αντιρρήσεις για περίπου 55% των περιπτώσεων ε, πάντα για το διοξείδιο του αζότου. Για το αξίδια, συγγνώμη, του αζότου. Από το Δεκέμβριο του 2012 μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2013 θα πάρουμε απόφαση για τις υπόλοιπε υποθέσεις για τη Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία και Λουξεμβούργο δηλαδή για κάποιες ζώνες αυτών των χωρών. Η Κομισιόν δέχεται ότι τα κράτη-μέλη ε, μπορούν να ζητήσουν ε, επέκταση για το οξύδιο του αζότου εφόσον φέρουν νέα στοιχεία που σύμφωνα με αυτά ε, το άρθρο 22 της οδηγίας του 850 θα γίνεται σεβαστό. Όλες οι λεπτομέρειες για τις ε, κοινοποίησεις και τις αποφάσεις ε, υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας. Προσπαθούμε λοιπόν να έχουμε μια διαφανή διαδικασία. Θα ξαναυποβληθούν στοιχεία, γιατί το επιτρέπουμε αυτό. Και αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε τη στρατηγική εφαρμογή, ειδικά για το διοξίδιο του άνθρακα και τα 10 ppm και θέλουμε να κλείσουμε ε, την αναθεώρηση του περιβαλλοντικού αέρα. Είμαστε δηλαδή εν μέσω μεταρρύθμισης, ας πούμε. Για το 10 PM έχουμε προσαγάγει 10 υποθέσεις στο δικαστήριο. Έχουμε τρεις αποφάσεις που έχουν εκδοθεί. Για τις υπόλοιπες εκκρεμίσεις υποθέσεις ετοιμάζουμε επίσημα σημειώματα για να εξασφαλίσουμε ότι τα απαραίτητα μέτρα θα ληφθούν ούτω ώστε να, οι υπερβάσεις να είναι στον πιο μη μικρές, όπως απαιτεί και η οδηγία. Με τα αυτά, κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί βουλευτές, νομίζω ότι σας έδωσα μία πλήρη εικόνα και σας απάντησα στις ερωτήσεις. Μπορώ να συμπληρώσω αν το επιθυμείτε. Αυτό είναι particles per something, έτσι. Ε, Σας ευχαριστώ. Όπως κατέστησα αφές φαίνεται πως γινόμαστε θύματα της επιτυχίας μας. Τα αυτοκίνητα γίνονται πιο καθαρά, αλλά με τις διάφορες τεχνολογίες ανέρχονται τα οξύδια του αζότου και βέβαια και λόγω της αύξησης αριθμού των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στα αστικά κέντρα. Είναι σωστό που τίθεται η ερώτηση σήμερα στην ημερήσια διάταξη, γιατί του χρόνου 2013 θα είναι το έτος του καθαρού αέρα και θα πρέπει κάποιες στρατηγικές να υιοθετηθούν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να καθαρίσει ο αέρας των πόλεων. Ο Βιτόριο Πρόντι έχει τώρα το λόγο και μετά η Λίντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Κομισιόν, για την απάντηση. Με, μετά από αυτά που ακούστηκαν πριν, να σας πω ότι στη ΣΤΟΑ έγινε μια μελέτη για την τοξικότητα των νανοσωματιδίων σε αιώρηση. Και όπως υπόθηκε, Ε, εκλείονται κυρίως από τους δίζελο κινητήρες. Το πρόβλημα νομίζω μπορεί να επιληθεί. Είναι ένα πρόβλημα των αστικών περιοχών. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο εξαρτάται από τις πηγές. Πού είναι οι κινητήρες εσωτερικής καύσης, κυρίως οι δίζελο κινητήρες όπως σας είπα και είπε και ο μιλητής της Κομισιόν. Περιμένοντας λοιπόν την ηλεκτρική έλξη, τους ηλεκτρικούς κινητήρες, όπου θα μας δω μια λύση, αν και όχι πλήρες, μπορούν να βοηθήσουν ε, ε, στο μεταξύ να βοηθήσει ας πούμε το μεθάνιο, ε, το φυσικό αέριο ως καύσιμο. Εγώ έχω ένα τέτοιο αυτοκίνητο και δεν εκλείω καθόλου σωματίδια. Τουλάχιστον αυτό το θέμα έχει εν επιληθεί. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να δώσουμε κίνητρα προς αυτήν την κατεύθυνση με το μεθάνιο κτλ. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Ούτε το πρόβλημα του διοξιδίου του αζότου. Εάν δεν δράσουμε σε επίπεδο πηγών που εκλείουν τα σωματίδια αυτά. Ε, πιο μακροπρόθεσμα η λύση είναι τα ηλεκτρικά οχήματα βέβαια η 100% ηλεκτρική έλξη. Αλλά αυτά είναι του μέλλοντος. Στο μεταξύ πρέπει να εμπιστευτούμε καύσιμα, διαφορετικά καύσιμα όμως, με την κατάλληλη χρήση, χρησιμοποιώντας τα σημερινά μέσα κίνησης που έχουμε. Yeah, I just wanted, um, Ευχαριστώ. Έχουμε το πρόβλημα της κυκλοφορίας, αλλά δεν είμαι σίγουρη. Έχουμε κάνει πρόοδο στο σχεδιασμό, ας πούμε, των αυτοκινήτων. Μπορούν οι τοπικές αρχές να σεβαστούν αυτά τα όρια η κατάσταση του στόλου των, των αυτοκινήτων και του θορύβου στην Ευρώπη. Ε, το λαμβάνετε υπόψη Κομισιόν. Κοιτάτε τα άλλα νομοθετήματα τα οποία υπάρχουν, μήπως δεν έχουν προχωρήσει αρκετά γρήγορα όσο έπρεπε. Λέτε ότι ξεκινάτε κάποιες διαδικασίες επί παραβάση, για να το καταλάβω καλά. Πώς εντάσσετε αυτό στην αναθεώρησή σας. Ξεκινάτε τις ε, διαδικασίες επί παραβάση πριν μεταρρυθμίσετε την νομοθεσία. Κομισιόν Να προσπαθήσω να είμαι ακριβή Καταρχάς, για την κυκλοφορία και για αυτά που υπόθηκαν σχετικά. Υπάρχει ένα αναφυσβήτο πρόβλημα Δηλαδή, οι, πραγματικέ οι πραγματικές εκπομπές. Υπάρχει μια έγκριση τύπου στα οχήματα που υποτίθεται ότι θα πρέπει να οδηγήσει σε πραγματική μείωση των ρηπογών ουσιών, των ορούμενων σωματιδίων δηλαδή και του διοξιδίου του αζότου. Το Euro 5, το Euro 5 που ισχύει, ε, μας λύνει εν μέρη το πρόβλημα ε, των αιωρούμενων ε, σωματιδίων. Είμαστε σχεδόν στην άκρη του τούνελ. Αλλά όμως έχουμε το πρόβλημα, το εξετάζουμε, το ψάχνουμε. Οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, συγγνώμη του αζότου, ε, ξεπερνούν πολύ το τι μπορεί να επιλύσει η έγκριση τύπου οχημάτων. Γιατί αν θυμάμαι καλά, οι εκπομπές, οι οριακές τιμές εκπομπών θα πρέπει να, ληφθούν, να θεσπιστούν λαμβάνοντας υπόψη τις ε, συνήθεις συνθήκες κυκλοφορίας, οδήγησης κτλ. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δηλαδή. Το θέμα δεν είναι να υπάρχει λοιπόν νέα νομοθεσία μόνο. Έχουμε καταλάβει πάντως ότι χρειαζόμαστε το Euro 6 και πρέπει να τεθεί θυμάστε το συντομότερο δυνατό σε ισχύ, γιατί το Euro 5 μας οδήγησε σε κάποια ε, φίλτρα για τα αιωρούμενα σωματίδια. Προσπαθούμε να τα παγιδεύσουμε λοιπόν. Και βλέπουμε ότι στο μεταξύ το μερίδιο του διοξιδίου του άνθρακα στο συνολικό μείγμα οξυδίων του αζότου αυξάνεται. Θα πρέπει υποτίθεται το Euro 6 να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Μπορεί το Euro 6 να μην αντιμετωπίσει συνολικά το πρόβλημα των, της μόλυνσης, γιατί το θέμα είναι τι επιτρέπουμε αυτή υπερβαίνει την πρόθεση του νόμου. Υπάρχουν διάφορα άλλα θέματα τα οποία πρέπει να αποφασιστούν και να αντιμετωπιστούν. Αλλά από ό,τι μας λέει και ο κλάδος, το Euro 6 θα μας δώσει τέλεια φίλτρα και επεξεργασία ε, της μόλυνσης και των ρηπογόνων ουσιών σε όλα τα οχήματα. Και μετά από αυτά που είπε, τα πολύ ωραία που είπε, αυτός ο, που είπε ο κύριος Πρόντι, Αυτά τα φίλτρα θα παγιδεύουν τους περισσότερους ρυπαντές, ακόμα και τα νάνο σωματίδια. Υπάρχουν διάφορα στοιχεία, κυρίως οι εξατμίσεις ε, των δίζελοκινητήρων που μας απασχολούν. Το θέμα είναι σε ποιο βαθμό οι κατασκευαστές θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν συστήματα διαχείρισης ε, ε, του κινητήρα μόνο και μόνο για να αποφύγουν ας πούμε τις συσκευές ε, επεξεργασίας που είναι πιο ακριβές. Μόνο αντιμετωπίσουμε τις πραγματικές εκπομπές θα διευκολύνουμε τις αστικές αρχές για να εφαρμόσουν τις οριακές τιμές εκπομπών. Όλα αυτά τα λέω με κάθε επιφύλαξη όμως, γιατί η μεταρρύθμιση δεν έχει η αναθεώρηση μάλλον δεν έχει ολοκληρωθεί, η επικύρωση κτλ. Αλλά σε σχέση με την ε, ποιότητα του αέρα υπάρχουν και κάποια θέματα διαχείρισης. Υπάρχει μια... Ε, απ' τη μία υπάρχουν ας πούμε οι ευθύνε των αρχών. Συχνά άλλα μας λένε οι τοπικές αρχές, άλλα οι εθνικές αρχές. Νομίζω ότι πρέπει να επιβάλλουμε, να προτείνουμε μάλλον εμείς, ε, πιο αυστηρή νομοθεσία που αφορά τις πηγές των ρηπαντών. Αυτό σε ένα πρώτο επίπεδο και μετά μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα υπόλοιπα με την αναθεώρηση. Τελευταίο. Δεν ξεκινάμε κατά ανάγκη διαδικασίε επί παραβάση πριν ολοκληρώσουμε την αναθεώρηση τη νομοθεσία. Γιατί καταρχά πρέπει να δούμε για ποια νομοθεσία, ποια είναι η πιο κατάλληλη νομοθεσία που πρέπει να, να υποβάλουμε για και ποιες νέες πρωτοβουλίες. Δεν πρέπει να είμαστε προθύστεροι. Πρέπει να κάνουμε μια πολύ σοβαρή ανάλυση πριν από αυτό. Είδαμε όμως ότι η εφαρμογή των πολιτικών έχει δρομολογήσει κάποια πράγματα, κάποιες δράσεις. Μερικές φορές γίνονται συζητήσεις, ας πούμε, δημόσιες. Και τα λέω με κάθε σεβασμό. Πάντως, για τις οριακές τιμές εκπομπών έχουμε βάλει, τις έχουμε βάλει στα τέλη της δεκαετίας 90, πολλά χρόνια πριν. Στην πραγματικότητα όμως αυτό που διαπιστώνω ότι συμβαίνει είναι ότι υπάρχει πολλή χαρτούρα, γραφειοκρατία κτλ. και λίγη δράση. Μπορούμε, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υποστηρίξουμε ε, τις δράσεις, τις όποιες δράσεις αναλαμβάνονται επιτόπου, με κάθε σεβασμό προς την επικουρικότητα. Αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις προτάσεις που θα υποβάλει η Κομισιόν του χρόνου. Παρακαλώ να επιταχύνετε την όλη διαδικασία έτσι ώστε να μας υποβληθεί εγκαίρως η πρόταση και να μπορέσουμε να την επεξεργαστούμε μέσα στην παρούσα θητεία. Σε ό,τι αφορά τα αυτοκίνητα οχήματα υπάρχει και ένα μεγάλο κενό μεταξύ θεωρητικών εκπομπών και εκπομπών στην πράξη. Πρέπει εδώ να εξετάσουμε και τι γίνεται με, τα, με τους κύκλους των τεστ, των δοκιμασιών αυτών των αυτοκινήτων στους οποίους ε, διαπιστώνονται ε, οι εκπομπές με τον τρόπο που γίνονται οι μετρήσεις προκύπτουν κάποια πλονεκτήματα υπέρ των κατασκευαστών. Η προσπάθεια που γίνεται να μειωθεί το διοξείδιο του ανθράκα συνολικά θα συμβάλλει και στην μείωση των εκπομπών των ε, καυσερίων. Έχουμε πολλούς πρώιμους, πρόωρους θανάτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, από ε, τέτοιες πηγές. 10 έως 15.000 ιδίως από τα οξύδια του αζότου. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλες και όλους όσοι συμμετέσχετε στη συζήτηση και για τις παρεμβάσεις σας, καθώς και την κυρία Μακάβαν για την ερώτηση. Θέλετε πάλι το λόγο? Ορίστε. Πολύ σύντομα γιατί Μόλις τώρα συνειδητοποίησα ότι δεν απάντησα στο θέμα του χρονοδιαγράμματος. Καταρχήν, μάλλον θα ολοκληρώσουμε τον Σεπτέμβριο και θα είναι πολύ δύσκολο να ε, επιταχύνουμε. Κυρίως ήθελα πάντως να σας πληροφορήσω ότι μπορείτε να παρακολουθείτε την επικείμενη ανάλυση και όλα τα σχετικά στην ιστοσελίδα μας. Μάλιστα σήμερα ή αύριο θα αναρτήσουμε τα τελευταία δεδομένα των σεναρίων της μέγιστης ε, δυνατότητας εφαρμογής, εφαρμοσιμότητας. Ευχαριστώ. Η συμβουλή μου είναι να, να δώσετε στους αυτούς σας χρόνο μέχρι το Σεπτέμβριο 2013. Αν μείνετε όμως μέχρι το 2013 τότε το Κοινοβούλιο δεν μπορεί πλέον δεν θα προλάβει πλέον το Κοινοβούλιο. Θα είναι πάρα πολύ κρίμα εάν η διαδικασία αυτή δεν μπορέσει να ολοκληρωθεί. Γι' αυτό κάντε κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιταχύνετε την διαδικασία. Μιλάμε, λέω ξανά ότι του χρόνου θα είναι το έτος του καθαρού αέρα. Είναι σκόπιμο το σημαντικό αυτό θέμα να ξαναμπεί στην ατζέντα για να μπορέσουν να ληφθούν και αποφάσει. Δεν έχει κανένα νόημα. Εάν δώσετε στον, στον εαυτό σα χρόνο μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2014, δεν πρόκειται πλέον το Κοινοβούλιο να προλάβει να το συζητήσει. Ευχαριστώ και εύχομαι καλό μεσημεριανό διάλειμμα σε όλου. Για το απόγευμα βρέστε και άλλου να έρθουν για να είναι γεμάτη η αίθουσα. Θα έχουμε ενδιαφέροντα θέματα.